Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα, συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Καλώς σας καλωσορίζω στην συνεδρίαση της ε, Φορολογικής Επιτροπής μας. Θα ήθελα να ξεκινήσει η σημερινή ακρόαση ως εξής. Αύριο θα συμπληρώσουμε ένα έτος από την δολοφονία της ε, Δάφνης ε, Γκαλίτσια της Μαλτέζας ε, δημοσιογράφου, την οποία είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πολλά μέλη της Επιτροπής Διαρρυθμίσεως των Panama Papers και θα ήθελα να τηρηθεί ενός λεπτού σίγη προς τιμή ε, τη κυρία Γαλίτσια και των άλλων δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν πρόσφατα και τη κυρία Μαρινόβα στην Βουλγαρία. Well, Όπως ξέρετε, η σημερινή συνεδρίαση αφορά μία ακρόαση για τις χρυσές βίζες και διάφορα άλλα τέτοια συστήματα φορολογικών προνομίων και θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα για τους κινδύνους ξεπλήματος χρήματος, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που σχετίζονται με αυτά τα προγράμματα. Και μετά θα μιλήσουμε για τις ελεύθερες οικονομικές ε, ζώνες, ειδικά αυτές ε, που λειτουργούν ως χώροι υποθήκευσης για αγαθά υψηλή αξίας, που είναι γνωστές γενικά ως ελεύθεροι λιμένες. Μετά ε, θα έχουμε λοιπόν δύο πάνελ. Το ένα θα ασχοληθεί με τις χρυσές βίζες, το άλλο με τις ελεύθερες λιμένες. Το πρώτο, στο πρώτο έχουμε καλέσει εκπροσωπούς του ΩΣΑ και της ΜΚΟ Global Witness και έχουμε εκπροσώπους της Κομισιόν από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης που θα απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις που θα τους απευθύνεται. Επίσης καλέσαμε τον διευθυντή της Πορτογαλικής Υπηρεσίας Μεταναστεύσεως και Συνόρων που διαχειρίζεται και το θέμα χρυσής βίζας, αλλά δυστυχώς ε, αρνήθηκε. Δεν ε, προσήλθε, οπότε δεν θα μπορέσουμε να ακούσουμε την άποψη του πορτογαλικού κράτους ε, που πιθανώς να έχει κάποια αιτιολόγηση για το σύστημα αυτό ή για να απαντήσει σε ερωτήσει των βουλευτών. Λοιπόν, όλοι οι βουλευτέ ε, έχουν λάβει τις γραπτές απαντήσεις. Ε, και βεβαίω είναι διαθέσιμες και στη σελίδα της Επιτροπής μας μετά την συνεδρίαση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πάνελ ε, κίνδυνοι στον τομέα του ξεπλήματος ε, χρήματος. Ε, να δούμε λοιπόν τους πρώτους μιλητές. Έχουμε τον κύριο Φίλιπ Κέρφς, επικεφαλής της Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας του ΟΣΑ. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Ραχίλ Όουενς, επικεφαλής της, των επαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οργάνωση Global Witness. Καλωσορίζω και την κυρία Βασιλιάδου, η οποία είναι τμήματάρχη του τμήματο ε, οικονομικού εγκλήματος στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη και την κυρία Μόνικα Μόσχαμερ, ε, η οποία επίσης είναι τμήματάρχη ε, για τα δικαιώματα των πολιτών και την ελεύθερη μετακίνηση από την ίδια Γενική Διεύθυνση. Ξέρετε πως έχουμε κάνει ήδη μια διαβούλευση για να μην γίνεται κατάχρηση αυτών των συστημάτων για να παρακάμπτονται τα κοινά, οι κοινές αναφοράς και βεβαίως θέλαμε ο κύριος Κέρφς να μας πει ποια είναι τα ευρήματα αυτής της διαβούλευσης αν και πιθανώς ε, τα ευρήματα αυτά να είναι προσωρινά και βεβαίως η οργάνωση Global Witness έχει εκπονήσει και μία μελέτη για τους κινδύνους αυτών των προγραμμάτων, οπότε θέλουμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Λοιπόν, θα εργαστούμε ως εξής. Ο κάθε μιλητής θα έχει 10 λεπτά να κάνει κάποιες παρατηρήσεις και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους βουλευτές. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τον κύριο Κέρφς να κάνει τις πρώτες του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σαν όσα, ως όσα. Αυτά τα προγράμματα επένδυσης δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε μεμονωμένα, αλλά το κάνουμε στα πλαίσια ενός συνολικότερου προγράμματος. Βέβαια ασχοληθήκαμε με τα θέματα αυτά, θα έλεγα κάπως επεισοδιακά. Στα πλαίσια των πληροφοριών που αρχίσαμε να συλλέγουμε, να γνωστοποιούνται αν θέλετε από την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πιστοτικών πληροφοριών ή πληροφοριών για καταθέσεις κτλ. και εκεί μπορούν τα κράτη να συλλέγουν πληροφορίες ε, από τα πιστοτικά τους ιδρύματα για τους μη μονίμους κατοίκους ε, των χωρών. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν έχει προχωρήσει αρκετά. Είχαμε μέχρι τώρα 102 ε, δικαιοδοσίες, εθνικές οι οποίες πήραν μέρος. Το πρώτο εξάμεινο του 17 ε, ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος θα έλεγα ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών και τον προηγούμενο μήνα ξεκινήσαμε για τα στοιχεία τα οποία συνελέγησαν στις αρχές του 2018. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει προχωρήσει λοιπόν στα πλαίσια του λεγόμενου After Sale Service σε εισαγωγικά Προσπαθούμε εμείς να δούμε σε ποιο βαθμό οι ρυθμίσεις ε, δεν εφαρμόζονται με τον προσήκοντα τρόπο και προσπαθούμε να δούμε ε, μέσω των πληροφοριών τις οποίες συλλέγουμε πού θα μπορούσαν να ανοίξουν παραθυράκια σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν έτσι ώστε να αποτρέψουμε στο μέλλον την παραβίαση των κανόνων. Και ακριβώς εκεί συναντήσαμε ε, την ιστορία αυτή με τις χρυσές βίζες. Οργανώσαμε στην αρχή του 18 γύρω από το φαινόμενο αυτό μία διαβούλευση. Συνεργαστήκαμε με διάφορες χώρες έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε σε ποιο βαθμό τα προγράμματα αυτά μπορούν να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης στα πλαίσια του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών. Έχουμε συμφωνήσει ήδη σε τεχνικό επίπεδο ορισμένα κριτήρια επί τη βάση των οποίων τα προγράμματα αυτά απόκτησης ε, άδεια παραμονής ε, με βάση την επένδυση ε, του συγκεκριμένου πολίτη μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο. Είναι δύο βασικά τα κριτήρια τα οποία εφαρμόζουμε. Το πρώτο is that the scheme should uh, only Καταρχάς, ε, τα ελάχιστα ε, ποσοστά, τα ελάχιστα απαιτούμενα ποσοστά φυσικής παρουσίας είναι το ένα κριτήριο και το δεύτερο βλέπουμε το επίπεδο φορολογίας το οποίο επιβάλλεται ή την μη δυνατότητα, ή την δυνατότητα μάλλον μη επιβολής φορολογίας ανάλογα με τις ρυθμίσεις οι οποίες επικρατούν σε κάθε χώρα. Βλέπουμε αν υπάρχει ας πούμε ένα γενικότερο καθολικό καθεστώς επιβολής φορολογίας, ε, σε ποιο βαθμό υπάρχουν δυνατότητες αποκλήσεων, εξαιρέσεων, και σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρξουν εκπτώσεις φορολογικές ή και πλήρεις απαλλαγές εφόσον έχει οργανωθεί ένα συγκεκριμένο σύστημα φορολογίας ή καλύτερα μη φορολογίας για τέτοιου είδους εξωτερικούς επενδυτές. Λοιπόν, χοντρικά θα είναι τα δύο κριτήρια, φυσική παρουσία από τη μία, φορολογία από την άλλη. Προσπαθήσαμε να δούμε ακριβώς αν θα μπορούσαν να βρεθούν αντίμετρα στην περίπτωση κατά την οποία σαν παράδειγμα υπάρχει άμεση ανταλλαγή πληροφοριών με την αρχική χώρα προέλευσης του επενδυτή και ένας άλλος παράγων μετρίασης του κινδύνου είναι η τεκμηρίωση η οποία θα πρέπει να απαρέχεται από τον υποψήφιο για την απόκτηση να πρέπει να είναι ε, επαρκής Σε σχέση λοιπόν με τα κριτήρια αυτά τα οποία προανέφερα, βρήκαμε τουλάχιστον 100 προγράμματα απόκτησης άδειας παραμονής μέσω επενδύσεων από το εξωτερικό. Υπάρχουν πολύ περισσότερα, δεν έχουμε καλύψει όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες από τις χώρες αυτές ε, υπόκεινται στην υποχρεωτική εφαρμογή του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις καταθέσεις των μη εγκατεστημένο στη χώρα. Και υπάρχει ένα ποσοστό των προγραμμάτων αυτών τα οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου σε σχέση με τη δυνατότητα αποφυγής εφαρμογής των κανόνων οι οποίοι είναι ενισχύ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δημοσιοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα υψηλού κινδύνου, όχι για να δακτυλοδείξουμε τις χώρες αυτές, αλλά για να δώσουμε τη δυνατότητα στα πιστοτικά ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα κοινό σύστημα, ένα τυποποιημένο κοινό σύστημα παρουσίασης και δημοσιοποίησης των στοιχείων, να τους δώσουμε όλα τα στοιχεία λοιπόν τα οποία απαιτούνται έτσι ώστε να μπορέσουν να φροντίσουν τα συμφέροντα του πιστοτικού του ιδρύματος και να χρησιμοποιήσουν όλες τις ε, δυνατότητες ενημέρωσης οι οποίες είναι διαθέσιμες. Και σε σχέση με το φορολογικό ε, για την συγκεκριμένη χώρα, αλλά και για φορολογικές επιβαρύνσεις και στις χώρες προέλευσης, γιατί και εκεί θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ε, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ανταλλαγή στοιχείων ανάμεσα στα πιστοτικά ιδρύματα της χώρας προέλευσης και της χώρας κατάληξης ε, του εμβάσματος προς επένδυση. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιες από τις χώρες ε, έχουν ε, δεχθεί να ξεκινήσουν εθελοντικά αυθόρμητα θα έλεγα την διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων, κάτι το οποίο αυτόματα θα μειώσει τον κίνδυνο ο οποίος ε, παρουσιάζεται από την εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων. Ε, εδώ βρισκόμαστε χοντρικά. Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσουμε σύντομα την διαδικασία στον όσα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σωστά και τις υπόλοιπες χώρες εκτός των 102 με τις οποίες είμαστε σε επικοινωνία. Αυτά. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ η κυρία Owens. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή Tax 3 που με προσεκάλεσε σήμερα να μιλήσω για τους κινδύνους διαφθοράς που έχουν σχέση με τα προγράμματα χρυσών θεωρήσεων, χρυσών βίζα. Ε, Είμαι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Global Witness και έχουμε επί 25 χρόνια προσπαθήσει να αποκαλύψουμε ε, υποθέσεις διαφθοράς. Πρώτα, για τα έσοδα από φυσικούς πόρους, όπως Καμπότζη, που φτάνουν σε ιδιωτικέ τσέπες. Σιγά σιγά αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει συστημική συμπεριφορά διαφθοράς και εμείς το αποκαλούμε αυτό κύκλος ζωής της διαφθοράς. Κλέβουν, αποθηκεύουν, δαπανούν. Αυτή, αυτά τα τρία ρήματα τι κλέβουν. Για παράδειγμα, ε, εδάφη που ανήκουν σε μια κοινότητα ανθρώπων ή ε, το τροπικό δάσος. Μετά αυτά τα μετατρέπουν σε χρήματα. Τα χρήματα αυτά μπορεί να τα αποθέτουν σε τράπεζες ή σε offshore και ε, μετά έρχονται να τα ταπανίσουν. στις περισσότερες περιπτώσεις αγοράζοντας εκλογές και πατρονάροντας πολιτικούς για να διατηρήσουν την εξουσία. Μετά από αυτά στρέφουν την προσοχή τους, οι κλεπτοκράτες δηλαδή, σε υψηλή αξίας αγαθά. Και εκεί έρχονται και οι χρυσέ θεωρήσει, οι χρυσέ βίζε που γίνονται πολύ ελκυστικέ, διότι μπορούν να αγοράσουν την ηθαγένεια ή το δικαίωμα διαμονή σε άλλη χώρα. Είναι μεν δαπανηρή υπόθεση, αλλά αποτελεί επένδυση, διότι δίνει στον ε, διαφθαρμένο ε, επιχειρηματία ή και στην οικογένειά του ε, τη δυνατότητα να ξεφύγει από τα ραντάρ των αρχών, να αλλάζουν τόπους, χώρες να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμού αλλού κλπ. Δεν εκπλαγήκαμε λοιπόν όταν πέρσι η εφημερίδα Guardian μαζί με έναν αριθμό δημοσιογράφων ξε, ξέθαψαν τέτοιες υποθέσεις διαφθοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη με επικεφαλής επιχειρήσεων όπου εμπλέκονταν και συγγενείς πολιτικών της Αγγόλα Ουκρανοί και ε, Ρώσοι ολιγάρχες οι οποίοι είχαν αγοράσει το δικαίωμα διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Πορτογαλίας και Κύπρου. Έχουμε συντάξει έκθεση όπου εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για το γεγονός ότι οι χρυσές θεωρήσεις που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν πλέον έμφυτο χαρακτηριστικό όλου του κύκλου διαφθοράς και ενισχύουν του ε, διεφθαρμένου επιχειρηματίε, προσφέροντά του ασφαλέ λιμάνι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έρευνέ μα δείχνουν ότι η διαχείριση των συστημάτων αυτών, κακή διαχείριση των συστημάτων, έχουν εκθέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τεράστιο αριθμό τέτοιων χρυσών θεωρήσεων που έχουν ύποπτα χαρακτηριστικά με συγκρούσει συμφερόντων κ.ο.κ. Για παράδειγμα, βρήκαμε ότι εξ όσων φαίνεται Κύπρος και Πορτογαλία δεν εξετάζουν την πηγή του πλούτου όταν εξετάζουν τις ε, αιτήσει για, χρυσή, ε, για χρυσές θεωρήσεις. Στην Άρτα επίσης, οι αξιωματούχοι έχουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια για την επιλεξιμότητα του ετούντος. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ποινικά μητρώα φορτωμένα και παρόλα αυτά υπό ιδιαίτερε συνθήκε μπορούν να γίνουν αποδεκτοί για χρυσέ θεωρήσει. Και πέρα από αυτά βεβαίω, έτσι φτάνουν αυτοί στην Ευρώπη, η ανάλυση μα δείχνει ότι η περιορισμένη λογοδοσία και διαφάνεια οδηγούν και σε αύξηση διαφθορά και μέσα στι ίδιε τι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα διακριτική ευχέρεια και πολύ χαμηλό ε, έλεγχο. Εμεί ασχολούμαστε με τα πράγματα αυτά από δύο πτυχέ. Πρώτον, θεωρούμε ότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. Όλοι οι ετούντε θα πρέπει να περνούν με τη δέωσα επιμέλεια από αυστηρότητα τους ελέγχους και να αναζητούνται οι συγκρούσει συμφερόντων η νομιμότητα της αιτήσεως πρέπει να επαληθεύεται και το background να ελέγχεται αυστηρά. Δεύτερο, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν την πεποίθηση ότι τα συστήματα αυτά ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ε, ασφαλείας και δεν επιτρέπεται να το παραβλέπουν αυτό οι κυβερνήσεις. Εδώ διαφάνεια και λογοδοσία είναι τα κλειδιά. Είναι κρίσιμο επίσης οι κυβερνήσεις οι οποίες επιλέγουν να προωθήσουν τέτοια προγράμματα να αρχίσουν ανοιχτό διάλογο με τους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί και η Ένωση και οι επιμέλους χώρες μέλη πρέπει να πούν και αυτές τι θεωρούν αποδεκτό. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να εξηγήσουν την επιχειρηματολογία υπέρ των συστημάτων αυτών και να διεξαχθεί ανοιχτή συζήτηση για τα λεγόμενα δίθεν ωφελήματα από τα συστήματα αυτά. Αυτό είναι κρίσιμο για την ασφάλεια κάθε χώρας μέλους αλλά και για την ακαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρε που προσφέρουν χρυσέ θεωρήσει να μην ταλίζονται από το αναμενόμενο κέρδο και λησμονούν την ανάγκη άσκηση δέουσα επιμέλεια ή αν έχουν δείξει δέουσα επιμέλεια, τελικώ να απορρίπτουν τα αποτελέσματα τη έρευνα αυτή. Και αυτά αφορούν ιδίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχουν οι κανόνε τη ελεύθερη κυκλοφορία, που σημαίνει ότι η απόφαση που λαμβάνει μια χώρα μέλο επηρεάζει όχι μόνο του δικού τη πολίτε, αλλά τεράστιες είναι, ε, είναι τεράστια επιρροή και για τη ζωή των υπόλοιπων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ξεκινά το σύστημα από εκεί. Παίρνετε ένα διαβατήριο, ενώ δεν χρειάζεται να έχετε 27. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες μέλη που προσφέρουν τέτοια συστήματα, στην ουσία εκμεταλλεύονται μια ευκαιρία για την οποία πληρώνουν οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. οι οποίες δεν ε, υποφελούνται ωστόσο από κανένα από τα λεγόμενα ωφελήματα. Ελεύθερη κυκλοφορία, εναρμόνιση προτύπων κλπ. στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί προστίθεται ακόμα ένα επίπεδο κινδύνου, διότι τα πρότυπα κατεβαίνουν προς τα κάτω και επομένως και η ιδέως επιμέλεια και ακαιρεότητα πάσχουν. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα, Η μεγάλη ελκυστικότητα της χρυσή ε, θεώρησης είναι ότι επιτρέπει ελεύθερη διακίνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς σύνορα και ε, βεβαίω ακόμη περισσότερο όταν ε, φέρνει και την ηθαγένεια. Και γι' αυτό αιτιολογείται, κατά τη γνώμη μας, να ληφθεί δράση σε επίπεδο ένωσης. Χαιρόμαστε την πρωτοβουλία της κυρίας Ιούροβα, η οποία δήλωσε ότι, τον Αύγουστο ήδη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται να γίνει ασφαλές λιμάνι για παράνομες δραστηριότητες και εγκληματίες. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι συγκεκριμένε δράσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει ένα αριθμό πραγμάτων. Πρώτα, για την τις επόμενες κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχει μια σειρά κριτηριών μεταξύ αυτών η διαφάνεια για τα συστήματα παραγωγή χρυσή θεώρηση. Να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτε γνωρίζουν του κινδύνου και τα λεγόμενα ωφελήματα από τα συστήματα αυτά. Να υπάρξει σχετική νομοθεσία και να υπάρξουν και μέτρα μετριασμού. Ενδεχομένω με ένα υπερεθνικό έλεγχο που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε λίγα χρόνια. Τρίτο, να προσθεθούν και απαιτήσει κατά της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Τέταρτο, να δημιουργηθούν μηχανισμοί για την διάδοση των πληροφοριών για να αποφευθεί να μετακινούνται ανάμεσα στις διάφορες δικαιοδοσίες και Και τέλος, να υπάρξουν και διαδικασίες κατά χωρών μελών οι οποίες παραβιάζουν την, ε, ε, τις αρχές της συνεργασίας για τα συστήματα αυτά. Πολύ ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις. Thank you very much. Well, now... ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάει τώρα η συζήτηση με τους ε, βουλευτές. Οι ερωτήσεις θα γίνουν σε πέντα λεπτά, Ένα λεπτό για την ερώτηση, τέσσερα λεπτά για την απάντηση. Όπως είπα, ε, υπάρχει η δυνατότητα να ρωτήσετε και την Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν τέσσερις ομιλητές, αλλά θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να περιορίσετε τον αριθμό των ερωτήσεων. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν με τους συνεισηγητές ε, πρώτα απ' όλα από το ΕΛΚΟ, κύριος Λούντεκ Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, δεν ξέρω εάν θα απαντηθεί η ερώτησή μου. Λοιπόν, μάθαμε ότι περισσότερα από τα μισά κράτη-μέλη έχουν τέτοια συστήματα. Επίσης, από την διεθνή διαφάνεια μάθαμε ότι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για το θέμα του ξεπλήματος χρήματος. Υπάρχουν όμως δύο ζητήματα που με απασχολούν. Το ένα είναι κάπως αφηρημένο, είναι ένα θέμα αξιών, δηλαδή το τι αγοράζει το χρήμα. Ε, υποτίθεται ότι η Ευρώπη βασίζεται σε κάποιες αξίες οι οποίες κατά κανόνα δεν πολλούνται. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν το χρήμα πρέπει να κάνει διαφορά. Ίσως κάποιος να είναι λιγότερο πλούσιος, θέλει να έρθει στην Ευρώπη, να φτιάξει μια επιχείρηση και μετά να δημιουργήσει κάποια φοβερή προσθεμινέξη. αξία. Ενώ κάποιος ο οποίο ήρθε και πλήρωσε, ε, μόνο κόστος θα έχει για την οικονομία. Απορώ λοιπόν. Αλλά τέλο πάντων, μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση είναι η εξή. Σε ποιο βαθμό εξετάζει ο κόσμο την οικονομική πτυχή. Ε, Βεβαίω, ε, στον 21ο αιώνα δεν νομίζω να υπάρχει ε, κάποια ε, έλλειψη κεφαλαίου, αλλά δεν μας λείπουν γενικώ οι επενδύσεις. Μας λείπουν οι επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και δουλειές ε, και ευημερία για την κοινωνία. Και ακριβώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε αυτά τα συστήματα, το ότι κάποιος δηλαδή αγοράζει ακίνητα ε, πολυτελή, ε, μπορεί πράγματι να δημιουργεί κάποια προσθέμενη αξία, αλλά κατά τα άλλα είναι μόνο κόστος για την οικονομία, δεν υπάρχει προσθέμενη αξία, μόνο ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων. Και αναρωτιέμαι ποια είναι η θετική πτυχή για την οικονομία. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια λογική, κάποιο ο οποίο έρχεται με τα λεφτά και λέει δώστε μου μια άδεια παραμονή και θα επενδύσω. Ε, Μήπω είναι κάτι του 1950 και δεν έχει θέση στον 21ο. Σα ευχαριστώ. Βεβαίω, φαντάζομαι υπάρχουν διαφορέ από το ένα σύστημα στο άλλο. Ποιο θα ήθελε όμω να απαντήσει. Ναι, κυρία Όμεν. Σα ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Ε, πραγματι είναι πολύ σωστά αυτά τα οποία αναφέρετε. Κατά την άποψή μας υπάρχουν πολλοί και βουλευτές παραδείγματος χάρη που λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι ο κίνδυνος διαφθοράς. Ένα τεράστιο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα εν λόγω κράτη-μέλη που επιτρέπουν δηλαδή να μπαίνουν τα άτομα αυτά στη χώρα και νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει πολλά και διάφορα από όλες τις ε, πλευρές ε, του ζητήματος. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο πολλών δισεκατομμυρίων. Φέρνει λεφτά στα κράτη-μέλη, αλλά το βασικό είναι ότι δεν ξέρουμε πόσα. Υπάρχει πλήρης έλλειψη διαφάνειας και έλλειψη διαφάνειας ε, για το τι γίνεται όταν μπουν αυτά τα λεφτά στα κράτη-μέλη. Υπάρχει πράγματι και ένα φαινόμενο που κάποια πολύ μικρά κράτη-μέλη αναζητούσαν έσοδα μετά την κρίση, αλλά αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ακριβώς ότι έχουμε έναν τέτοιο ανταγωνισμό. Ε, δηλαδή, μπροστά στα κέρδη κλείνουν τα μάτια στο τι φέρνουν αυτά τα άτομα. Ε, γιατί είναι οικονομική πτυχή οπωσδήποτε θα το εξετάσει οπωσδήποτε η Επιτροπή σας ποια είναι τα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη ε, των ε, συστημάτων αυτών και αν υπάρχουν τέτοια, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη διαφάνειας. Εμείς ε, τέσσερις μήνες γράφουμε αυτή την έκθεση, δεν υπάρχει καθόλου δημόσια πληροφόρηση και είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια αξιολόγηση για το εάν αυτά τα πράγματα είναι καλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να προσθέσει κάτι. Κύριε Κέρβς, να πω συγκεκριμένα ότι στο επίπεδο του ΩΣΑ δεν έχουμε κοιτάξει τα συγκεκριμένα αυτά συστήματα εξ όσων γνωρίζω για ζητήματα ξεπλήματος χρήματος ε, ούτε την ηθική πτυχή του φαινομένου και ε, πόσο ξέρω δεν έχουμε εξετάσει και το σκεπτικό των χωρών όταν κάνουν κάτι τέτοιο. Τι σκοπεύουν να πετύχουν οι χώρες ε, μακροπρόθεσμα. Μπορεί να κάνουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Ο Σάσαφος ε, έχει πείρα από παράλογες ε, κινήσεις ε, διαφόρων κρατών. Ευχαριστώ Κόφωτ, σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και <coughs> το πάνελ μας. Επιτρέψατε μου να επαναλάβω κάποιους αριθμούς από την διεθνή διαφάνεια. Τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 100.000 άδειες και διαβατήρια έχουν εκδηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα αυτά, όχι μόνο σε μία χώρα, αλλά στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 25 δις άμεσες επενδύσεις αλλά δυστυχώς μόνο δύο χώρες έχουν δημοσιεύσει πλήρη στοιχεία για τις ξένες επενδύσεις, τα υπόλοιπα δεν είναι ιδιαίτερα διαθέσιμα. Είστε πεπισμένοι ότι τα προγράμματα αυτά βασίζονται σε πραγματικού τύπου επενδύσεις και σε πραγματική συμμετοχή στην οικονομία των χωρών. Το ΩΣΑ έχει εξετάσει την υπόθεση αυτή ότι υπάρχει πλήρης μεταφορά πόρων στις νέες οικονομικές δικαιοδοσίες. Ε, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι προσωπικοί οικονομικοί λόγοι που οδηγούν σε αυτή την επένδυση. Και δεύτερον, μπορείτε να αναφερθείτε σε ένα τέτοιο τουλάχιστον πρόγραμμα το οποίο εσείς θεωρείτε ότι είναι βέβαιο και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για πλήσιμο βρώμικου χρήματος. Θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο. και πιστεύετε ότι ε, τα προγράμματα τα οποία έχετε εξετάσει σε μία χώρα μήπως υπάρχει ουσιαστική μεταφορά των προγραμμάτων αυτών στις επόμενες χώρες. ο εκπρόσωπος του ΩΣΑ. Κοιτάξτε, εμείς το εξετάσαμε αυτό στα πλαίσια μιας στενής προοπτικής, θα έλεγα. Είδαμε ότι υπάρχει μια τρομακτική ποικιλία για τέτοιου είδους προγράμματα, από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια προγράμματα όπου δεν υπάρχει καμία, κανένα αντικείμενο πραγματικής επένδυσης, απά πρέπει να υπάρξει πληρωμή. Και υπάρχουν προγράμματα τα οποία είναι διαφορετικά και λειτουργούν στα πλαίσια της προσέλκυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Υπάρχουν λοιπόν τα δύο άκρα. Αυτά τα οποία έχουμε εξετάσει εμείς είναι θα έλεγα αυτά τα οποία μπορεί να μην είναι πραγματικές επενδύσεις. Εμείς βέβαια το εξετάζουμε αυτό στα πλαίσια της κατάχρησης και της αγνόησης των ε, κανόνων που είναι ενισχύ. Αν δει και τα κριτήρια αυτά κανείς, μόνο αυτά τα κριτήρια, αν και υπάρχουν και άλλα, τότε μπορεί να πει ότι υπάρχουν ε, ορισμένα από τα προγράμματα αυτά τα οποία πράγματι δεν παρουσιάζουν κινδύνους. Αν κάποιος θέλει ας πούμε να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα στο Βέλγιο για να αποκτήσει ε, άδεια παραμονής, είναι μια χώρα η οποία έχει υψηλά φορολογικά επίπεδα, υψηλά ποσοστά επιβολής, οπότε ε, είναι κάτι το οποίο δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο ενώ υπάρχουν άλλες χώρες ε, οι οποίες θα εξυπηρετούσαν πολύ καλύτερα τους στόχους ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν την φορολογία και χώρες οι οποίες ε, δεν απαιτούν να γνωστοποιούνται τα προσωπικά οικονομικά στοιχεία αυτού ο οποίος καταθέτει ε, ένα συγκεκριμένο ποσό. Η κυρία Owens. Εγώ δεν πρόκειται να κρίνω αυτή τη στιγμή το κάθε ένα από τα προγράμματα αυτά. Εμείς προσπαθούμε να ασχοληθούμε με θέματα διαφθοράς και κατάχρησης ε, των ε, κανόνων. Τώρα, σχετικά με το αν είναι μια επένδυση, πραγματική επένδυση. Βλέπουμε την κατάσταση στην Πορτογαλία, βλέπουμε να υπάρχουν πάρα πολλά ποσά χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε ακίνητα, στρεβλώνουν την αγορά ακινήτων της συγκεκριμένης χώρας σε ορισμένες περιοχές και είναι προγράμματα βέβαια τα οποία λειτουργούν σε σχέση με ε, την κάλυψη των συμφερόντων των επενδυτών. Βέβαια υπάρχει μια ουσιαστική έλλειψη γνώσης της προέλευσης ε, των ποσών αυτών. Ε, πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία είναι πλήρως ελεύθερη θα έλεγα, δεν διακανονίζεται με κάποιον τρόπο. Όλοι οι άλλοι τομείς, ε, είτε μικροί είτε μεγάλοι, ελέγχονται και διακανονίζονται. Ένα άλλο σημείο η ουγγρική περίπτωση, το ουγγρικό παράδειγμα, έχει επιβεβαιωθεί σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί το ουγγρικό πρόγραμμα. Στο παρελθόν η κατάσταση ήταν τέτοια όπου το κράτος έχανε ουσιαστικά από το πρόγραμμα αυτό γιατί τα επιτόκια για τα κρατικά ομόλογα τα οποία θα έπρεπε να προσπαθήσουν να αποκτήσουν οι επενδυτές, αυτές, οι επενδυτές αυτοί για να πάρουν την άδεια ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία πλήρωνε η ίδια η Ουγγαρία για τα χρήματα τα οποία δανειζόταν σαν χώρα. Οπότε εκεί δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης του επιχειρήματος αυτού σε σχέση με την το οικονομικό κέρδος το οποίο θα μπορούσε να έχει. Κάτι αντίστοιχο είχαμε στη Βουλγαρία Είχαμε το παράδειγμα όπου η τράπεζα της Βουλγαρίας, μια επενδυτική κεντρική τράπεζα στη Βουλγαρία, έδινε δάνεια ε, σε ξένους επενδυτές έτσι ώστε να τα επενδύσουν τα χρήματα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. Υπάρχουν κάποιες περίπλοκες καταστάσεις, όπως επίσης υπάρχει το θέμα των τιμών στις οποίες πολλούνται τα ακίνητα και σε ποιο βαθμό θέτουν σε κίνδυνο την ισορροπία της αγοράς. Κοιτάξτε, ε, δεν ζήτησαν όλες οι πολιτικές ομάδες το λόγο. Θα ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αν θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Ε, η κυρία Γκόμες. Όταν πήγαν τα έγγραφα του Παναμά στην χώρα μου, την Πορτογαλία, δηλαδή σε εξεταστική επιτροπή, είχαμε πολλές ερωτήσεις. Λίγα όμως μάθαμε για το πρόγραμμα αυτό. Και βεβαίω για την προέλευση των κεφαλαίων που έφερναν οι ενδιαφερόμενοι. Τώρα στην Πορτογαλία, από τον Οκτώβριο του 2012, πάνω από 6.000 θεωρήσεις έχουν χορηγηθεί και πάνω από 11.000 άνθρωποι κατόρθωσαν να έρθουν στα πλαίσια της επανένωσης οικογενειών Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να ειδεί κανεί την σύμπτωση των χωρών των ετούντων. Κινέζοι είναι οι περισσότεροι στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Δεν επιτρέπεται να φέρουν πάνω από 50.000 Τώρα, για να αγοράσει κανεί ένα κινητό στην Πορτογαλία για να αποκτήσει τη χρυσή βίζα, πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον 350.000 ευρώ. Και αυτά ανοίγουν οδού έλευση του οργανωμένου εγκλήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν της διαφθοράς. Είναι λοιπόν πραγματικά παράξενο που ο ΣΑΡΑ δεν έχει ακόμη ενδιαφερθεί, διότι μιλώ πράγματι για μια μείωση των προτύπων μεταξύ των χωρών μελών, δηλαδή έναν ανταγωνισμό προς τα κάτω, που θα μπορούσε να θεωρηθεί και παράνομη ε, κρατική ε, επιδότηση, προς το οργανωμένο έγκλημα στην πραγματικότητα, αλλά και βεβαίως και σημαντική κίνδυνη ασφάλειας, ιδίως για ορισμένες χώρες όπως Μάλτα και Κύπρο, όπου Αυτό που κάνουν είναι να διαφημίζουν την δυνατότητα διέλευσης των συνόρων Σέγγεν όταν δίνονται αυτές οι χρυσές βίζες. Και κάποιος μου είπε τελευταία ότι αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν μπορούν πλέον να απελαθούν, δεν μάλλον εκδοθούν στην περίπτωση που πρέπει να δικαστούν στις χώρες τους ως εγκληματίες. Και τώρα, ποια είναι η γνώμη σας για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με τις χώρες μέλη για να οργανώσουν τέτοια λεγόμενα δίθεν εισαγωγικών επενδυτικά προγράμματα. Και στην περίπτωση της Μάλτας είδαμε ε, μια συγκεκριμένη επιχείρηση που έπαιξε ένα ιδιαίτερα ιταμό ρόλο και μιλήσαμε προηγουμένως, μάλλον ε, ε, ε, ε θυμηθήκαμε προηγουμένως την επέτειο της του θανάτου της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίσια, η οποία δολοφονήθηκε λόγω του ότι αποκάλυψε τις ε, ιστορίες αυτές και βεβαίω όσα είχε πει τότε η δημοσιογράφος ήταν αλήθεια για την επιχείρηση αυτή. Υπάρχουν και, άλλες, και άλλοι όμιλοι με τους οποίους μάλιστα παρευρέθηκε και ο ίδιος ο ο πρώην, πρώην ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε επαφές με το Μαυροβούνιο και με άλλους. Βέβαια και οι μεγάλοι τέσσερις φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο σε παρόμοια προγράμματα. Η πτυχή της ασφάλειας πώς είναι δυνατόν να αγνοείται συστηματικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όχι μόνο από τις χώρες μέλη που ε, τους επιτρέπεται να αναπτύσσουν αυτά τα ε, ποταπά προγράμματα. Ας απαντήσει πρώτη η κυρία Όουενς στην ερώτηση της κυρίας Γκόμες. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Είπα κάτι προηγουμένως. Πρόκειται για μια ολόκληρη βιομηχανία που δεν είναι ρυθμισμένη αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να καλυφθεί από τους κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος, γιατί συχνά ο ρόλος που παίζουν είναι να διαχειρίζονται τεράστια ποσά και να τα ξεπλύνουν και ε, ε, ελεύθεροι από οποιαδήποτε, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδους νομοθετική ρύθμιση. Και σωστό είναι αυτό που είπατε, ότι ο CEO, το Hennen Partners, αποκλήθηκε ο βασιλιάς των διαφατηρίων. Και έχει παίξει όντως τον ρόλο αυτό να κάνει δηλαδή τις άδειε διαμονής και διαβατήρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πολυτελές αγαθό. Πολλοί θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ τα διαβατήριά της στον, στην υψηλότερη προσφορά χωρίς να κάνει απολύτως κανέναν έλεγχο. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η νομοθετική ρύθμιση. Θεωρώ επίσης ότι υπάρχει και κάποια ανησυχία σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων όπως είπατε πριν, για την υπόθεση της Μάλτας, όπου η εταιρεία Henian Partner όχι μόνο προσελκύουν τους ε, επενδυτές αυτούς, αλλά κάνουν και τον έλεγχο. Και στην περίπτωση των Κινέζων επενδυτών, για παράδειγμα. Ο άλλος κίνδυνος είναι η προσπάθεια να είναι επιτυχής οι αιτήσει, δηλαδή μια επιχείρηση η οποία λαμβάνει χρήματα για να περνά μέσα από το σύστημα περισσότερου ετούντε, αυτό είναι βεβαίω ένα κίνητρο για την επιχείρηση αυτή να αυξήσει τον αριθμό των ετούντων και να κλείσει επομένως ένα και δύο μάτια απέναντι στους κινδύνους διαφθοράς. Όπως είπε και η κυρία Γκόμε, πρόκειται για μια τεράστια βιομηχανία πηγαίνετε για διακοπές στην Κύπρο και βλέπετε τεράστιες διαφημίσεις για τα προγράμματα αυτά, για αυτούς που φτάνουν στα κυπριακά αεροδρόμια. Τους δίνετε κάθε είδους πληροφορία για τις προσφορές που κάνουν οι επιχειρήσεις αυτές και νομίζω ότι όντως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να εγκύψουν να δουν περί τίνος πρόκειται και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που συνεπάγεται όλη αυτή η υπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς και Κέρφς, αλλά παρακαλώ σύντομα. Φέρατε εκεί πέρα δύο μεγάλους παίκτες σε αυτή την υπόθεση και υπάρχουν και πολύ μικρότεροι. Είχαμε συζητήσεις με αυτούς και εντός του κλάδου υπάρχει θα έλεγα μια αντίληψη ότι χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Δεν ξέρω αν ο σκοπός είναι ο ανταγωνισμός ή να σταματήσουν τον ανταγωνισμό αλλά είναι σαφές ότι η ρύθμιση του κλάδου έχει κάποια ωφέλη αν ε, δεν ανησυχεί ε, πολύ κανείς ε, για την νομοποίηση της ίδιας της έννοιας ε, της παροχής άδειας παραμονής μεσοπενδύσεων. Αλλά βεβαίως θα οδηγήσει σε περισσότερη επιμέλεια σε όλους τους τομείς και στον τομέα που με αφορά, την φορολογία δηλαδή, ναι, γιατί βεβαίω θα πρέπει να υπάρχουν ε, σωστές ε, διαδικασίες δίουσας επιμέλεια, έτσι ώστε η υπηρεσία που ασχολείται με την αίτηση να μπορεί να βρει την πραγματική ε, χώρα κατοικίας του ετούτος. Οπότε υπάρχουν κάποια ωφέλη. Σας ευχαριστώ από την Κομισιόν, η κυρία Μόσχαμα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω λίγο το τι κάνει και η Κομισιόν. Κατόπιν του Κοινοβουλίου Μάλιστα. Απεξεργαζόμαστε μία έκθεση και αξιολογούμε τα συστήματα αυτά ε, και για την άδεια παραμονής και για τις ε, υπηκότητες γιατί συχνά τα βάζουμε σε ένα τσουβάλι. Θα δούμε λοιπόν ε, και τα δύο συστήματα αυτά και συνεργαστήκαμε με έναν εξωτερικό συνεργάτη για να αναλύσουμε την νομική κατάσταση και ελπίζουμε να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τον οικονομικό αντίκτυπο αλλά είναι κάπως δύσκολο να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Ακόμα το επεξεργαζόμαστε οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για μια τελική εξελόγηση. Επίσης προφανώς συντάσσουμε και την έκθεση Οπότε δεν μπορώ να σας πω τώρα κάτι συγκεκριμένο για το τι κατευθύνσεις θα δοθούν. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία αναφέρθηκαν ε, ζητήματα και τρομοκρατίας, ε, ξεπλήματος χρήματος, ε, φόρο διαφυγής, όλα αυτά τα οποία έδεσαν. Και χαιρόμαστε που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον ΩΣΑ γιατί βεβαίως και η έκθεση της ε, διεθνούς ε, διαφάνειας οπωσδήποτε είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στην έκθεσή μας, την οποία θα υποβάλουμε πριν το τέλος του έτους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από το ECR υπάρχει κάποιος. Όχι. Συλλελεύθερος. Ναι, Βολφ Κλίντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ λόγω του Brexit Υπάρχει μια αύξηση των πολιτών οι οποίοι θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρώπης των 27 και πάρα πολλοί εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν να πάρουν την Βρετανική υπηκότητα. Θεωρείται ότι αυτή η κατάσταση χρησιμοποιείται και για να υπάρξει δυνατότητα απόκρυψης ε, και χρήσης χρημάτων τα οποία έχουν ε, κερδιθεί με παράνομο τρόπο εκτός του κανονικού επίσημου πιστοτικού δικτύου. Εφόσον υπάρχει μια δημόσια διοίκηση η οποία σέβεται ε, το νόμο και προσπαθεί να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις που ισχύουν. Έχουμε στοιχεία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στους ε, παράνομους, τους εγκληματικούς κύκλους και στη δημόσια διοίκηση ή σε εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης. Τι στοιχεία έχετε γύρω από αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση. Σχετικά με τις επενδύσεις σε ακίνητα. Εγώ ζω στο Βερολίνο και τα τελευταία 4-5 χρόνια οι τιμές των ακινήτων έχουν πραγματικά πάει πάρα πολύ ψηλά και οι επενδυτές προέρχονται από χώρες όπου δεν φαντάζεται κανείς ότι υπάρχουν πλούσιοι επενδυτές, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία κτλ. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των επενδύσεων προφανώς χρησιμοποιούνται για να πληθεί βρώμικο χρήμα. Νομίζω ότι η απλή ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών ανάμεσα στις ε, γερμανικές ας πούμε αρχές που συλλέγει ε, τον φόρο απόκτησης ακινήτου και που πρέπει να ενημερώνει τις ε, χώρες από τις οποίες προέρχεται η επένδυση. Κάποιος που στέλνει χρήματα από την Αθήνα στο Βερολίνο για να αγοράσει ένα πολυτελές διαμέρισμα πρέπει να είναι σίγουρος από ό,τι φαίνεται ότι δεν ενημερώνεται η Αθήνα για τη συγκεκριμένη αγορά. Κυρία Ούντς. Εγώ μπορώ να απαντήσω στον τομέα στον οποίο έχω την δυνατότητα να το κάνω. Για τα ακίνητα. Εμείς ε, σε συνεργασία και με εταίρους όπως με την Transparency International προσπαθούμε να υπάρχει ε, μεγαλύτερη διαφάνεια και το ίδιο γίνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γίνεται μία προσπάθεια για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων και να προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από τις επιχειρήσεις ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και επενδυτές. έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επενδύουν, ιδιαίτερα στον τομέα των ακινήτων. Είδαμε ότι υπάρχει ένα σύστημα ουσιαστικής απόκρισης των πραγματικών ιδιοκτητών. Αυτό είναι ο βασικός στόχος λοιπόν, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε σωστά το από πού προέρχεται η επένδυση. Τώρα για το Brexit δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να, για το οποίο μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα το τι θα γίνει. Αυτό το οποίο λέμε και πολλές ΜΚΟ ζητούν είναι να ισχύσουν οι ίδιοι όροι και οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση για το πλήσιμο του βρώμικου χρήματος. και η οδηγία η σχετική με το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις έτσι ώστε να εφαρμόσουν σωστά τις νομοθεσίες που επιτρέπουν την δημοσιοποίηση της πραγματικής επιχείρησης που φέρεται ως ιδιοκτήτρια και υπάρχει φόβος ότι μετά το Brexit τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν θα γίνουν σεβαστές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιες τέτοιες ενδείξεις θεωρείται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει ε, με τους ίδιους περίπου κανόνες. Ευχαριστώ. Η πράσινη. Να συνεχίσω αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Νίντεμάγερ. Η ιδιότητα, αν θέλετε, η υπηκότητα μπορεί να είναι ένα απλό εμπόρευμα το οποίο πωλείται και αγοράζεται. Μήπως ε, δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει δυνατότητα αγοράς ουσιαστικά. Έχουμε αρκετές ε, πληροφορίες ε, σχετικά με το πλήσιμο του βρώμικου χρήματος μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα και είναι απαράδεκτο το ότι υπάρχουν χώρες που το δέχονται. Θα ήθελα επίσης να μάθω αν έχετε πληροφορίες για τις απάτες που γίνονται στο εσωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για Ιταλούς, για Γάλλους, οι οποίοι αγοράζουν βουλγαρική υπηκότητα ή υπηκότητα της Μάλτας ή αυστριακή υπηκότητα, κυπριακή υπηκότητα, για να αποκρύψουν ακριβώς την πραγματική του ταυτότητα και να αποφύγουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την χώρα προέλευσης. Υπάρχουν από ό,τι φαίνεται αρκετά παραθυράκια σε σχέση με το σύστημα υποχρεωτικής ανταλλαγής. Ε, φαίνεται ουσιαστικά ότι είναι εύκολο να κάνει κανείς κάτι τέτοιο ε, Πραγματικά στην ουσία μπορεί να ανοίξει κανείς λογαριασμούς offshore με την ε, νέα ιδιότητα πολίτη, με τη νέα υπηκότητα την οποία έχει αγοράσει. Και δεν ξέρω αν έχετε επιπλέον στοιχεία και από τη Γαλλία ε, σε σχέση με το πόσο σημαντική είναι ε, η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα σε μια χώρα σαν τη δική μου. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε σχέση με τους νέους κανονισμούς, αλλά ίσως να μην είναι καν απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο. Για το δεύτερο θέμα, έχετε, αν έχουμε παραδείγματα, δεν έχω στοιχεία, αλλά όπως ε, είπαμε υπάρχουν διάφορα παραθυράκια. Είμαστε σε επαφή με και όλα και ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, δικηγόρους και τα λοιπά. Και μας έχουν, έχουν πλησιάσει διαφορετικοί γόροι που λένε ότι τα συστήματα αυτά διαφημίζονται, προωθούνται. Έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα ευρωπαϊκό κράτος που διαφήμιζε την υπόθεση αυτή στο Μεξικό, σε Μεξικανούς πολίτες. δεν ξέρω τις διαστάσεις που έχει. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για συγκεκριμένους αριθμούς. Περισσότερο ανεκτολογικά είναι τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ, κυρία Όνς. Δυστυχώς και εγώ την ίδια απάντηση έχω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπε και η Κομισιόν, να βρούμε πληροφορίε για τις ε, ροές εντός της ε, Ένωσης και συμφωνώ μαζί σας ε, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουν τα θεσμικά όργανα και πάλι για τα κονδύλια η αίσθηση που έχουμε είναι ότι δεν είναι ένα από τα χειρότερα συστήματα συστήματα όσον αφορά την έλλειψη ακεραιότητας και διαφάνειας αλλά ήταν και πάλι δύσκολο να βρούμε κάποιες προφορίες. Οπότε οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε με τα κράτη-μέλη για περισσότερη διαφάνεια θα μας βοηθούσε. Και για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα, συμφωνώ πλήρως μαζί σας και νομίζω ότι ένας από τους στόχους ε, της οργάνωσής μας ήταν ακριβώς να γίνει αυτή η συζήτηση. Και δεν έχουμε καταλήξει ε, στο εάν πρέπει να απαγορευτούν ή όχι, γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι τέτοιο χωρίς περισσότερες προφορίες. Όπως είπα, επί τέσσερις μήνες προσπαθούσαμε να βρούμε μια ανάκρη και ακόμα δεν ξέρουμε πώς ε, λειτουργεί αυτή η υπόθεση, αλλά οπωσδήποτε νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα εν ώψη των ευρωεκλογών που οι ευρωβουλευτές ε, και τα κράτη-μέλη πρέπει να ρωτήσουν τους πολίτες. Θέλουμε να πουλάμε την άδεια παραμονής ε, και την υπηκότητα. Ε, χωρίς διαφάνεια βεβαίως δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ είναι κανείς. Όχι. Η FTD. Η NF. Όχι κύριε Όχι. Το ΙΕΝΕΦ, όχι. Το ΕΛΚ. Και ο Σνίτερμαγερ. Να κάνω άλλη μία ερώτηση. Για το θέμα αυτό έχουν εντύπωση πως ε, τα κράτη δεν έχουν κάποιο οικονομικό σκεπτικό. Γιατί ειλικρινά το ότι κάποιος ε, έχει αγοράσει κάποια κρατικά ομόλογα χωρίς να... Δεν οφείλει αυτό μια χώρα τον 21ο αιώνα. Το ίδιο και αν αγοράσει ένα πολυτελές ακίνητο ή και αν επενδύσει σε μια εταιρεία που μπορεί να έχει εκατοντάδες διαφορετικούς ε, μετόχους. Ε, θεωρείται ότι δεν υπάρχει άρα κάποια ουσιαστική οικονομική ανάλυση των αποφάσεων αυτών που είναι κάτι το οποίο απλά είναι μια συνήθεια από το παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Mm. Νομίζω ότι η κατάσταση διαφέρει. Υπάρχουν ε, πολλά μικρά νησιωτικά κράτη εκτός Ευρώπης όπου ίσως να μην έχουν κάποια ξεκάθαρη στρατηγική πέρα από το ότι χρειάζονται το εισόδημα και ζουν μόνο από τον τουρισμό και αυτό είναι άλλη μια πηγή εισοδήματος και έχουμε άλλες χώρες, ε, μεγάλες χώρες έχουν κάποια συστήματα που προσπαθούν να προσελκύσουν επενδυτές στην χώρα. Αλλά ενδιαφέρον θα ήταν να το δούμε έτσι από κοντά. Και τους δύο τύπους αυτούς ε, συστημάτων. Και στις χώρες όπου η πρόθεση είναι να προσελκύσουν πραγματικούς επενδυτές ε, στις εταιρείες ε, με το τι προσπαθούν να επιτύχουν. Ε, εντάξει, είναι εκτός ε, το τομέα μου, αλλά προσωρινά θα ήταν προσωπικά με συγχωρείτε, θεωρώ ότι θα ήταν ενδιαφέρον να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ κυρία Όνης. Χαίρομαι που ακούω τόσα πολλά ερωτήματα για αυτό το θέμα γιατί η οργάνωσή μου θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι κατανοητό το ποια είναι τα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη. Τα νούμερα είναι σαφή βεβαίω. φέρνει χρήμα στις χώρες και έχουμε κάποια στοιχεία για κάποιες χώρες. Αλλά όπως σας είπα το μεγάλο θέμα είναι το πού πάνε αυτά τα λεφτά. Και επειδή δεν υπάρχει κάποια ακαιρεότητα, το ερώτημα είναι τι γίνεται, πάνε, τα τσεπώνει κάποιος υπάλληλος τα λεφτά αυτά και μετά εάν πάνε παραδείγματο χάρη σε ένα ταμείο στη Μάλτα υπάρχει ένα ταμείο κοινωνική ανάπτυξη όπου πάνε τα λεφτά αλλά μετά ακούσαμε ότι κάποια από αυτά τα χρήματα πηγαίνουν για να αγοράζουν μετοχέ σε τράπεζες δεν ξέρω αυτό αν ωφελεί του πολίτε τη Μάλτα ή του Ευρωπαίου πολίτε. και όσον αφορά τώρα το θέμα των κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά κράτη στην Καραϊβική που προσφέρουν αυτή τη στιγμή πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα. Έχουμε λοιπόν μια άλλη διάσταση εδώ. Δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, που έχουν αυτά τα συστήματα, αλλά και χώρες της Καραϊβικής, οι οποίες έχουν ε, πρόσβαση χωρίς βίζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσω της απαλλαγής που έχουν συμφωνήσει ε, η υπηκότητά τους είναι άλλος ένας τρόπος να έχει κάποιος ε, πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανώς και ένας διεφθαρμένος εγκληματίας. Είναι πολύ μικρά λοιπόν νησιωτικά κράτη, η Αντίγουα και η Μπαρμπούντα νομίζω όπου για να είναι κανείς ε, κάτοικος αρκεί να μένει πέντε μέρες ε, το έτος ε, και παίρνει μετά διαβατήριο και ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι ένα παραθυράκι θα έλεγα και βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν να πάει κανείς να παραλάβει το διαβατήριο. Το διεκπεραιώνουν κάποιες εταιρείε σου φέρνουν το διαβατήριο και μπορείς να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι άλλο ένα θέμα που πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εάν ξεκινήσουμε να μειώνουμε τους κινδύνους εντός της Ένωσης, υπάρχει και αυτό το παραθυράκι των χωρών εκτός Ένωσης που έχουν πρόσβαση στην Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιφάνος Περές. Κύριε Πρόεδρε, για την κυρία Όενς, στην έκθεσή σας μαζί με την ε, διεθνή διαφάνεια, κατά κάποιο τρόπο εκφράζεται μια επιφύλαξη ή μια κριτική απέναντι στην πέμπτη οδηγία κατά της νομοποίησης παρανόμων εσόδων, όπου μιλούμε για τις ε, υπόχρεες ε, οντότητες. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσχέρεια ανάθεσης μιας δημόσιας εξουσίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και το παράδοξο του νομοθέτου εν προκειμένου, από αυτό που καταλαβαίνω είναι μια πτυχή του θέματος που σας ανησυχεί. Έχετε άλλες προτάσεις που θα μας επέτρεπαν να επιλύσουμε το πρόβλημα. Δεν λέω ότι μπορούμε να να το προσθέσουμε στην δέσμη μέτρων που βρίσκονται ήδη επιτάπητος. Εγώ θέλω να καταλήξει η νομοθετική αυτή προσπάθεια. Αλλά μια και μιλούμε για την υπόθεση αυτή, καλό θα ήταν να είχαμε κάποιε κατευθύνσει από μέρου σα. Δεύτερο, για τον κύριο Κέρφ του ΟΟΣΑ. Σε μια από τι απαντήσει σα, είπατε ότι υπάρχουν 20 χώρε προβληματικέ. Μπορείτε να τι πείτε, ποιε είναι, ή εν πάση περιπτώσει να μα πείτε αν είναι κάποιε που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 ή των 27 ή της ζώνης ευρώ. Ευχαριστώ εσείς κύριε Κέρφης. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν σας έθεσα υπόψη τον κατάλογο είναι διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί απολύτως οι σχετικές εργασίες. Μπορώ να σας πω όμως ότι στην λίστα του προγράμματος αυτού που υπάρχουν χώρες που αποτελούν κίνδυνο, υπάρχουν και ορισμένες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες ΩΣΑ και κάποιες καραϊβικής. Ζώνη ευρώ, ρωτάτε. Νομίζω πως ναι. Παρατηρήσει χωρίς μικρόφωνο από την κυρία Μπέρες. Η κυρία Owens. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συνεργαζόμαστε, Global Witness και ε, διεθνή διαφάνεια και με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι ισχυρό το κείμενο της ε, οδηγίας κατά του ξεπλήματος του μαύρου χρήματος και για πρώτη φορά αποκαταστάθηκε ο σύνδεσμος, η διασύνδεση μεταξύ των χρυσών θεωρήσεων και της νομοποίησης παρανόμων εσόδων, του ξεπλήματος δηλαδή του μαύρου χρήματος. Από όσο ξέρουμε, υπάρχουν ωστόσο τόσα πολλά θέματα που χρειάστηκε να συμφωνηθούν στην οδηγία αυτή, που είμαστε ευγνώμονε που ξεκίνησε τουλάχιστον η πολιτική κατάσταση, ε, συζήτηση μάλλον και ανάλυση. Και εξετάζουμε τώρα ποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Η δική μας κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι είναι καλό μεν ότι η πέμπτη οδηγία AML αναφέρεται στον κίνδυνο που προέρχεται από τα προγράμματα χρυσών θεωρήσεων, αν όμως οι τράπεζες αναλάβουν και θέτουν τις ερωτήσεις, ρωτούν δηλαδή είστε ετών για χορήγηση ε, θεώρησης, Αυτό δεν αρκεί. Και πώ θα διασφαλιστεί ότι η πληροφορία θα περάσει από το πιστοτικό ίδρυμα, την τράπεζα κλπ. στην αρμόδια δημόσια αρχή τη χώρα μέλου Και ότι θα γίνει όντω η ανταλλαγή πληροφοριών. Και ποιο είναι υπεύθυνο εν τέλει για να αποφασίσει εάν ο ετών επιφέρει τον κίνδυνο του ξεπλήματος μαύρου χρήματος ή όχι. Και αν υπάρξει η πέμπτη οδηγία, θα πρέπει ενδεχομένως κάποτε να αναθεωρηθεί και για να αντιμετωπιστεί αυτή η βιομηχανία των χρυσών θεωρήσεων, η οποία πρέπει να καλυφθεί μέσα στους κανόνες αυτούς. Νομοθετικά δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπερέζη, αλλά χωρίς μικρόφωνο. Η κυρία Βασιλιάδου τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούστηκε συχνά η οδηγία για το ξέπλυμα μαύρου, μαύρου χρήματο. Και η ερώτηση τη κυρία μου δίνει αφορμή να πω ορισμένα πράγματα. Η οδηγία, να μην λησμονούμε τον στόχο τη, είναι προληπτικό εργαλείο. Να προλάβει δηλαδή την νομιμοποίηση του παράνομου χρήματο επιβάλλοντα υποχρεώσει για μια συγκεκριμένη συναλλαγή, όχι ένα γενικό και αόριστο κίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν εφόσον υπάρχουν ύποπτε συναλλαγέ θα πρέπει να κοινοποιούνται αυτέ τι αρμόδιε αρχέ, οι οποίε θα κάνουν κάποιου έλεγχου. Με την πέμπτη λοιπόν οδηγία, άλλωστε με πρωτοβολία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με σχετική τροπολογία τη κυρία Γκόμε, θεωρούμε ότι μπορούμε να περιλάβουμε τι χρυσέ βίζε. Αν πάει κάποιο λοιπόν σε μια τράπεζα να κάνει μια συναλλαγή και πρόκειται για πρόσωπο το οποίο θα ζητήσει χρυσή θεώρηση, πρέπει εκεί να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι. Εάν υπάρχει κάποια υποψία για το ποιόν τη συναλλαγή, θα πρέπει αυτή η υποψία να κοινοποιηθεί. Η κυρία Όεν είπε ότι καμιά φορά αυτό θα γίνεται εκ των υστέρων. Δηλαδή θα έχει δοθεί ήδη η θεώρηση και εκ των υστέρων θα γίνει ο έλεγχο. Δεν γίνονται πάντοτε οι έλεγχοι πριν από την επένδυση. Στι περιπτώσει αυτέ λοιπόν μπορεί να γίνουν εκ των υστέρων, αλλά μπορεί να γίνουν και από πριν. Η Rachel Owens λέει, λέει επίση ότι οι οντότητε οι οποίε διαχειρίζονται τα investment schemes θα πρέπει να γίνουν υπόχρεες οντότητε, obliged entities. Δεν είμαι απολύτω βεβαία, ότι, διότι η δική μας ανάλυση δεν μας επιτρέπει να είμαστε βέβαιε ότι αυτό είναι επαρκές, διότι η οδηγία, η πέμπτη οδηγία, εξετάζει συγκεκριμένες συναλλαγέ. Εάν λοιπόν η συγκεκριμένη συναλλαγή, στη βάση τη οποία κάποιο προσπαθεί να αποκτήσει τη χρυσή βίζα, προκαλεί κάποιε υποψίε, τότε ναι, σε ορισμένε περιπτώσει κάποιοι θα προσπαθούν να κάνουν επενδύσει και να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτε με χρήματα που είναι απολύτω καθαρά. Εκεί δεν θα προβληθεί υποψία. Δεν είμαστε λοιπόν βέβαιε ότι αυτό είναι το κατάλληλο εργαλείο. Η ίδια η Επίτροπος Γιούροβα είπε ότι χρειάζεται κάποια δέουσα επιμέλεια. Σε ορισμένε περιπτώσει θα είναι παρόμοια με αυτή που έχουμε στη Money Laundering Directive, αλλά ίσω η Money Laundering Directive να μην είναι το κατάλληλο όχημα. Μιλούμε επίσης πολύ για τράπεζες. Ως γνωρίζετε όμως, η οδηγία δεν αναφέρεται μόναχα στις τράπεζες. Εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο επιθυμεί να αγοράσει ακίνητη περιουσία, οι μεσίτες θα πρέπει να εξετάσουν αν υπάρχουν υπόνοιες. Το ίδιο απευθύνεται και σε δικηγόρους ή λογιστές, οι οποίοι χορηγούν συμβουλές σε αυτούς που υποβάλλουν αιτήσει για να γίνουν ε, πολίτες μιας χώρας μέλους. Είναι λοιπόν ένα συνολικό πλαίσιο για την ομοποίηση παρανόμων ε, εσόδων, αλλά για ειδικέ συγκεκριμένε συναλλαγές. Και να εξεταστεί, είναι ο ενδιαφερόμενος κάποιος ο οποίος ενδέχεται να ε, προσπαθεί να ξεπλύνει μαύρο χρήμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στη βάση γενική. Έχουμε τώρα αιτήσει για το σύστημα Catch VI, προσέλκυση της προσοχής του Πρόεδρου. Πρώτα η κυρία Γκόμες. Να υπενθυμίσω εδώ ένα σχετικό θέμα, το οποίο έθεσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ασαμινοτζάντ, Ιρανός πολίτης, ιδιοκτήτης της τράπεζας Πιλάτους, είναι λήφθης στις Ηνωμένε Πολιτείες και εννοώ την Πιλάτους στη Μάλτα, για παραβίαση της πιστοτικής νομοθεσίας και για πλήσιμο βρώμικου χρήματος. Είχε την δυνατότητα απόκτησης εγγράφων λειτουργίας στη Μάλτα το 2014 με διαβατήριο Saint Kitts and Nevis το οποίο του δόθηκε μέσω μιας συγκεκριμένης επιχειρήσης της Alien Partners, η οποία συναντάμε πολύ συχνά και πολλοί, πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ε, για ε, τέτοιες χορηγήσεις διαβατηρίου. Μας υποσχεθήκατε το Νοέμβριο την έκθεσή σας, πότε θα βγει. Εγώ θα συμφωνήσω με την Εύα Ζολή ότι η πώληση υπηκότητας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απαγορευθεί. Δεν είναι θέμα προσέλκυσης ε, ταλέντου ή επενδύσεων. Πόσο ταλέντο δεν πνίγεται στη Μεσόγειο αυτές τις μέρες. Αλλά το ελάχιστο θα ήταν να υπάρχει δημοσιοποίηση από πλευράς των κρατών μελών και κάποιες χώρες όπως η Μάλτα και η Κύπρος δημοσιοποιούν τα ονόματα. Η Κύπρος εκ των προτέρων, η Μάλτα ε, μαζί ανακατεμένοι με αυτούς που παίρνουν υπηκότητα για άλλους λόγους και αποκτούν την ιδιότητα του πολίτη της Μάλτας, αλλά άλλοι δεν το κάνουν και η δική μου χώρα δεν το κάνει. Και είμαι βέβαιος ότι ο μοναδικός λόγος που δεν το κάνουν δεν δίνουν ε, σε μένα είναι ότι φοβούνται ότι θα βρεθούν πάρα πολλά υποκείμενα εκεί τα οποία θα είναι πολύ αμφισβητήσιμα για να μην πω ε, εγκληματικής προέλευσης. Ευχαριστώ, Κομισιόν. Για το πότε, οπωσδήποτε πριν το τέλος του έτους ε, προσπαθούμε να κινηθούμε γρήγορα. Οπωσδήποτε πριν το τέλος του έτους για τα αιτήματα να απαγορευτεί εντελώς ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η απόδοση υπηκότητας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε προσεκτικά τις υποθέσεις. Έχουμε την περίπτωση Ρότμαν, την υπόθεση Ρότμαν και την υπόθεση Νότεμπομ επίσης ε, ε, Ενό διεθνού δικαστηρίου, διεθνούς δικαστηρίου απόφαση. Οπότε ε, είναι παρόλα αυτά αρμοδιότητα των κρατών και πρέπει να ε, έχουμε κατά νου αυτές τις πτυχές. Αλλά συμφωνώ μαζί σα ότι η διαφάνεια είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε ένα τέτοιο σύστημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ακούμε ότι οι ιδιωτικές τράπεζες σε κάποιες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν θέματα ασφαλείας δεν είναι πολύ ελκυστικές για επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επενδύσεις προς τέτοιου είδους πιστοτικά ιδρύματα. Το θέμα τι γίνεται με τις μεγάλες περιουσίες, τι γίνεται με τις επενδύσεις σε ακίνητα και τι γίνεται σε σχέση με την νομοθεσία του Σέγγεν και τους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι η Ντάφνε Καρουάνα είχε διερευνήσει και είχε καταγγείλει τις ελλείψεις σεβασμού ε, των κανόνων στη Μάλτα στα πλαίσια της ε, πώληση ουσιαστικά διαβατηρίων της Μάλτας και γι' αυτό και δολοφονήθηκε. Ε, όταν είχαμε έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι είχε ζητήσει μία μελέτη και στα πλαίσια της μελέτης φαινόταν ότι εφαρμόζονται ορισμένα κριτήρια να διασφαλίσουν την ασφάλεια της συναλλαγής ε, τα ελάχιστα επίπεδα χρόνου που πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε να γίνει η επαλήθευση των στοιχείων κτλ. Όμως στην ουσία βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν προγράμματα τα οποία διευρύνονται όλο και περισσότερο αντί να μειώνονται και να γίνονται πιο αυστηρά. Και εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω αν ε, αυτή τα, τα ευάλωτα χαρακτηριστικά του συστήματό μας ε, θα συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες τις οποίες κάνει σε αυτή την φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μία. Υπάρχει το θέμα ε, των ε, ακινήτων το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας δεν είναι υποχρεωτικά κάτι το οποίο συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες, αλλά υπάρχει το θέμα του βρώμικου χρήματος και της διαφθοράς, το οποίο διερευνούσε και η Τάφνε Καρουάνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την μελέτη στην οποία αναφέρθηκα στην πρώτη μου παρουσίαση, εμείς αναλύουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε διευρύνει την ανάλυση μας στις υπόλοιπες χώρες που, για τις οποίες δεν χρειάζεται βίζα. Συνειδητοποιούμε όμως την κατάσταση ε, που υπάρχει ότι οι κάτοχοι τέτοιου είδους ε, καθεστώτων, απελευθέρωσης των θεωρήσεων δηλαδή, ε, μπορούν να κυκλοφορούν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Και έχουμε και έναν τελευταίο γύρο, τον Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε δύο χρόνια το θέμα. Έχουμε εξεταστική επιτροπή και εδώ πέρα βέβαια η Κομισιόν θα έπρεπε να έχει υποβάλει μια πρόταση προκαιρού ε, για να τήρουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις στα κράτη-μέλη για την έκδοση βίζας ε, και τα λοιπά και επιπλέον ε, να επιδιώξουμε και μια ρύθμιση με τις τρίτες χώρες. Όπως είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, δεν αμφισβητείται ότι η απόδοση υπηκότητας είναι υπόθεση των κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε υπό ποιες συνθήκες ε, αποδίδεται η υπηκότητα. Γι' αυτό δεν βλέπω μία πρόταση της ε, Κομισιόν. Το θέμα είναι γνωστό. Δηλαδή το θέμα της ελάχιστης ε, παραμονής ή η ετήσια παρουσία ή κάποιο είδους τεστ που θα πρέπει να δίνει κάποιος η διάρκεια τη ε, επένδυση. Αυτά θα έπρεπε να ελέγχονται και να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο. Και μια απαγόρευση επίσης της επιθετικής αυτή διαφήμιση που έκανε παραδείγματο χάρη ο Πρωθυπουργό τη Μάλτας στο Χονγκ Κόνγκ. Όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία θα μπορούσε να κάνει μια λογική πρόταση η Κομισιόν χωρίς να αμφισβητεί το δικαίωμα των κρατών μελών. Και καλό θα ήταν να πάει ένας τέτοιο στην συναπόφαση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και όχι ότι πως γίνεται με τη φορολογία που απαιτείται ομοφωνία. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στα φορολογικά, του χάρη, πρέπει... Ε, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος θέλει στην ε, Γερμανία να εκμεταλλευτεί το γερμανικό ή το ελβετικό φορολογικό δικαίωμα παρά το ότι υπάρχει μια συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας, να έχει ένα ελάχιστο διάστημα παραμονής ε, στην χώρα. Γι' αυτό λοιπόν ε, το ερώτημα προς την Κομισιόν και τους ειδικού είναι το εξή ε, Έχετε κάποια ιδέα κατά νου για το πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο, γιατί ο χρόνος περνάει. Αν αφήσουμε και άλλα χρόνια να περάσουν δεν χρειάζεται να το συζητάμε άλλο. Yeah, commission. Ε, ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε, η Κομισιόν θα υποβάλει μια έκθεση αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ τώρα να σας πω τι θα περιέχει. Αλλά οπωσδήποτε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν εδώ και αλλού είναι πολύ σημαντικά και θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και Εύανση δεν ξέρω κάποιος άλλος. Ε, ήθελα να πω κι εγώ ε, ότι νομίζω ότι είναι προεκλογικό ζήτημα. έχουμε μήνες από τις ευρωεκλογέ και νομίζω ότι επαφείται στους βουλευτές να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τους ψηφοφόρους τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά και οπωσδήποτε αυτό θα βοηθήσει και από πλευράς πολιτικής βούλησης θα έχουμε άλλη κομισιόν του χρόνου και ελπίζω μετά το κοινοβούλιο αυτό να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση και να δημιουργηθεί ακριβώς πολιτική διάθεση για αλλαγή. έχουμε μια αλλαγή από το 2014 όταν ξεκίνησε το κοινοβούλιο να συζητά αυτό το θέμα. Ε, νομίζω ότι Πρέπει να ασκήσουν πίεση οι βουλευτέ. Ε, έχουμε νομίζω ξεπεράσει το εάν πρόκειται για ζήτημα Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ή όχι. Ε, το θέμα τώρα είναι πώς τα θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να βρουν μια λύση. Σα ΕΕ ευχαριστώ. Ωραία. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές σαφές ότι το ζήτημα αυτό είναι ένα θέμα φλέγων το οποίο γύρει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις και αναμένουμε την πρόταση της Κομισιόν και θα το παρακολουθεί το θέμα η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ τελείως εδώ το πρώτο μέρος της ε, συζήτησης. So colleagues, please take, take your seats. We will start another panel in a minute. Ξεκινάμε σε ένα λεπτό το επόμενο πάνελ. Ο πρόεδρος. Ας αρχίσουμε τώρα με το δεύτερο πάνελ Freeport, ειδικέ οικονομικές ζώνες, ευεργετήματα και κίνδυνοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω τους ομιλητές του δεύτερου πάνελ που είναι ο κύριος Πιεσάρντι από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Τσάρλ Καρ ε, ε, εμπειρογνώμων για χρηματοπιστωτικά. Καλώ ήρθατε. Ο κύριο Φαμπιέν Γκράσερ, δημοσιογράφος και συντάκτης του Le Quotidien και ο κύριο Κερμόντ που είναι διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση φορολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, τα πρόσωπα αυτά είναι διατηθειμένα να απαντήσουν σε ερωτήσεις όσο συνέβη και προηγουμένω η μέθοδος εργασίας θα είναι ίδια όπως και για το πρώτο πάνελ, δηλαδή τα α, τρία αυτά πρόσωπα θα έχουν λίγα λεπτά για να ε, κάνουν τις εισαγωγικές τους τοποθετήσεις και πρώτος ο κύριος Πιασάρδη για ε, να ε, κάνει την εισαγωγική του τοποθέτηση. Ορίστε παρακαλώ. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας προσφέρει να παρουσιάσουμε τη μελέτη που μας ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη χρηματοδότηση μάλιστα κιόλας μαζί με την ομάδα χωρών ΑΚΕ, την Ελβετική Κυβέρνηση, και την Ορβηγία και την Αυστρία. Η μελέτη αποτελεί μέρος του προγράμματος ε, ανταγωνιστικής βιομηχανίας και καινοτομία. Στην ουσία πρόκειται για ένα αναλυτικό έργο και σε επίπεδο χωρών και σε επίπεδο γνώσεως. Έχει ως σκοπό να δώσει νέα πνοή την εκβιομηχάνηση των αναπτυσσόμενων χωρών και των αναφιόμενων αγόρων. Έχουμε έως τώρα συλλέξει μελέτες από 36 χώρες και 6 knowledge products, προϊόντα γνώσεως. Ένα από αυτά είναι και για τις ειδικές οικονομικές ζώνες και μια επιχειρησιακή εξέταση των οικονομικών τους επιπτώσεων. Το πρόγραμμα έχει ανατεθεί σε ένα trust fund από την Παγκόσμια Τράπεζα και η μελέτη για τις ειδικές οικονομικές ζώνες αποτελεί μια εκτίμηση των πραγμάτων που απέδωσαν τα τελευταία 20 χρόνια σε προγράμματα και έργα της Παγκόσμιας Τράπεζας, ειδικώ για την ανάπτυξη των ειδικών οικονομικών ζωνών. Όταν αρχίζουμε μάλλον με έναν ορισμό, όταν μιλούμε δηλαδή για ειδικές οικονομικές ζώνες, αναφερόμαστε στην πραγματικότητα σε παραδοσιακές αλλά και υβριδικές export processing zones και για τις εξαγωγές επομένως και για τις εγχώριες αγορές. Μιλούμε επίσης για free port και δεν μιλούμε δηλαδή για ελεύθερο εμπόριο ούτε για ελευθερία του επιχειρήν. Δεν μιλούμε για τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα. Για να σας ε, δώσω κάποια νούμερα τώρα, βλέπουμε λόγω της παγκοσμιοποίησης αλλά και μετά ας πούμε από την ανάκαμψη της αγοράς μετά, μετά από το 2008-2009 βλέπουμε στο σημερινό κόσμο περίπου 3.500 ειδικέ οικονομικές ζώνες και τις υποδιαιρούμε σε ομάδες περίπου 120, λίγο πάνω από 120 χώρες με ειδικέ οικονομικές ζώνες. Βλέπει κανείς ότι έχουμε μια ταχεία αύξηση στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη. Τώρα το ε, ενιολογικό πλαίσιο, ο στόχος ήταν να διαπιστώσουμε τι, ποια πράγματα έχουν αποδώσει, ποια όχι, και τι θα πρέπει να μελετήσουμε. Βλέπουμε σύντομα ότι για να δημιουργηθεί η ειδική οικονομική ζώνη, πρώτα χρειάζεται ένα είδος δέσμης κινήτρων, δημοσιονομικών και μη δημοσιονομικών. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής χρειάζεται με κάποιο τρόπο να προσελκυστεί. Έχουμε μετά κάποιες, ε, κάποια σύνολα απαιτήσεων απαιτήσεων επενδυτικών, απαιτήσεων κυριότητας και μετά μπαίνουμε σε μια κατάσταση που έχει σχέση με τη διακυβέρνηση. Δηλαδή, πρωτίστως την ανεξαρτησία του ρυθμιστού και κυρίως η ρυθμιστική αρχή της ειδική οικονομικής ζώνης. Αυτή η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και βέβαια και το χρονοδιάγραμμα για την ε, τελική διαμόρφωση της ε, ελεύθερης ζώνη. Τώρα τα χαρακτηριστικά. Οριμότητα, μέγεθος, ε, διαχείριση, τόπος, industry focus, υποδομή, προσφερόμενες υπηρεσίες. Όταν μιλούμε για υποδομή θα πρέπει αυτό να το εννοήσουμε με ευρύτατους όρους, όχι μόνο πρόσβαση στο λιμάνι για παράδειγμα, αλλά πρέπει να δούμε επίσης και την παροχή ενέργειας, τις ε, ψηφιακέ υπηρεσίες, με την έννοια δηλαδή την ευρύτερη υποδομή. Έχουμε μετά τους ε, ε, περιβάλλοντες παράγοντες που έχουν σχέση με το πού τοποθετείται η ειδική οικονομική ζώνη. Έχουμε μετά και την θεσμική ποιότητα το κράτος δικαίου, την ε, πρόσβαση, την εγκύτητα στις αγορές, το επίπεδο εσόδων, το ανθρώπινο κεφάλαιο, αν είναι εκπαιδευμένο ή εκπαιδευμένο το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την πληθυσμιακή πυκνότητα. Στο επόμενο βήμα εξετάζει κανείς ποια από τα στοιχεία αυτά έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για τις ειδικέ οικονομικές ζώνες. Βλέπετε στο γράφημα ανάλυση που έχει γίνει για 207 ελεύθερες οικονομικές ζώνες και πρόκειται να προσθεθούν και ορισμένες ακόμη στο προσεχής μέλλον. Και πρώτα ας δούμε ότι έχουμε δημόσιες, ιδιωτικές ή μεικτού χαρακτήρα. Βλέπουμε πάντα από τη βάση δεδομένων ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο συνήθις στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική, ενώ η εμπλοκή του δημοσίου περισσότερο στην Ασία και στην Υποσαχάρη Αφρική. Βλέπουμε επίσης ιδιωτικό χαρακτήρα περισσότερο στην Κεντρική Ασία. Βλέπουμε ακόμη το χαρακτηριστικό του μεγέθους σε εκτάρια εδάφους. Στην υποσαχάρη Αφρική είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζώνες αυτές, μικρότερες Λατινική Αμερική και Καραϊβική. στη Κεντρική Ασία και Ασία βλέπουμε καμιά φορά και μεγαλύτερες ή μικρότερες και στη Νότια Ασία, δηλαδή στην Ινδία στην πραγματικότητα, εκεί χρειάζονται λιγότερο εμβαδόν, λιγότερο ε, ε, έδαφος. Αυτό προέκυψε από τη μελέτη, εν πάση περιπτώσει. Το, το, γράφημα είναι σημαντικό. Πρόκειται για τις εξαιρέσεις από την εταιρική φορολογία, που συμβαδίζει λίγο πολύ και με ε, το αντικείμενο της εργασίας σας και βλέπουμε ότι συνήθως βλέπουμε ότι πλησιάζουμε περισσότερο, ο μάλλον όσο πλησιάζουμε στην Ευρώπη, βλέπουμε λιγότερο από δεκαετία φορολογικών απαλλαγών, ενώ σε άλλες περιοχές είναι άνω της δεκαετίας. Βλέπουμε επίσης, εάν η ρυθμιστική αρχή είναι δημόσια αρχή, αν αυτή είναι απολύτως ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ότι στην Αφρική έχουμε μικτές αρχές, ενώ στην Ασία είναι πολύ πιο ανεξάρτητες οι ρυθμιστικές αρχές. Τώρα, η απόδοση. Δύσκολο να αναλύσει κανείς την απόδοση των ελεύθερων οικονομικών ζωνών, των ε, ειδικών οικονομικών ζωνών. Έχουμε ακόμα ε, εμπειρικά δεδομένα. Γίνονται φωτογραφίσεις άνωθεν των φωτισμένων χώρων τη νύχτα και βλέπει κανείς την επέκτασή τους ανά έτος. Έχουμε κάποιες που αυξάνονται, έναν αριθμό που μένουν ως, έμειναν, ε, ως, είχαν και έχουμε και συρρήκνωση. Όταν υπάρχει αύξηση σε πέντε χρόνια, από το 2007 έως το 2012, μιλούμε για μέση αύξηση της τάξης του 10%, ενώ η μέση αύξηση είναι μόνο 2,4%. Και, και βλέπουμε και μια ε, τυπική απόκληση του, της τάξης του 21% στην απόδοση. Αυτό δηλαδή δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε η ειδική οικονομική ζώνη θα αποβεί επιτυχής. Και στο πίνακα που βλέπετε τώρα δείχνουμε πώς θα πάνε. Έχουμε στην Νότια Αφρική πάλι 80% αύξηση, αλλά 20% συρρήκνωση. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που έχουν θετική επίπτωση, αρνητική επίπτωση ή δεν έχουν καμία συσχετισμό από την αρχή που θα γίνει μια επένδυση σε τέτοια ειδική οικονομική ζώνη. Οι εξαιρέσεις από την εταιρική φορολόγηση είναι ασφαλώς ένα ε, θετικό αποτέλεσμα η επιδότηση των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια που χρησιμοποιούν οι ε, οικονομικές ε, ζώνες, όπως για παράδειγμα το ρεύμα, επίσης. Έχουμε όμως και άλλα, δηλαδή ελάχιστη επένδυση, ε, διαδικασίες μοναδικής θηρίδας κλπ. Έχουν καμιά φορά επίπτωση και καμιά φορά όχι στην δημιουργία των ειδικών οικονομικών ζώνων. Έχουμε και δύο πράγματα τα οποία ε, είναι αντίθετα με την επενδυτική προσπάθεια. Αφενός τα έτη λειτουργίας, δηλαδή αν βρισκόμαστε προς το τέλος της περίοδου της επενδύσεως, αυτό μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην απόδοση της ειδική οικονομικής ζώνης. Και μετά η στόχευση στην υψηλή τεχνολογία, η οποία καθώς κινείται ταχύτατα, Πολύ συχνά μπορεί να συμβεί ότι είναι απερχαιωμένη πολύ σύντομα η τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Και τώρα οι περιβάλλοντε παράγοντε, Εκεί έχουμε περιβαλλοντικοί παράγοντε, Έχουμε ας πούμε την εγκύτητα σε μεγάλες αγορές. Αυτό ασφαλώς είναι θετικό. Εάν υπάρχει, αν μάλλον προϋπάρχει μια βιομηχανική βάση και αυτό είναι θετική επιπτώσεως, κάτι το οποίο διακόπτει ο πρόεδρος. Με συγχωρείτε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι, τελειώνω, τελειώνω. Και τέλος το περιφερειακό ε, κατακεφαλήν εισόδημα. ΑΕΠ μάλλον κατακεφαλήν, το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη επίπτωση για τις ειδικέ οικονομικές ζώνες. Αυτά είναι βασικά τα συμπεράσματα. Οι επενδυτές αναζητούν φθηνές τοποθεσίες με εγκύτητα σε μεγάλες αγορές αυτό είναι θετικό όπως είπα. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί απόδοση συν τον χρόνο. Υπάρχει η τεχνολογική συνιστόσα, επίσης και οι επιδοτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά δεν τα λέει η Κομισιόν, σημειώνω, αλλά η Παγκόσμια Τράπεζα σε μελέτη την οποία ανέθεσε. Σας ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και εγώ, κύριος Σκάρα. Ευχαριστώ, καλησπέρα σα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, όπως και το προηγούμενο. Τα ωφέλη και οι κίνδυνοι από μια οικονομική ένωση με και ζώνες ελευθερίου εμπορίου. Ακούσαμε κάποια πράγματα, κάποια άλλα ωφέλη που βλέπω εγώ. Προφανώς υπάρχει ε, ασφάλεια στα μέρη αυτά, ειδικά ο ελεύθερος λιμένας του Λουξεμβούργου και στην Γενέβη ε, υπάρχουν κάποιες ζώνες υψηλής αξίας, ελεύθεροι λιμένες, όπου φυλάσσονται κάποια προϊόντα υψηλή αξία. Υπάρχει λοιπόν το όφελο τη ασφάλεια, ε, βοηθά τι άμεσε ξένε επενδύσει, προωθεί το εμπόριο ε, και είναι αποτελεσματικό στον αφορά τη φορολογία, καταργεί διάφορου φραγμού και υπάρχει και ένα βαθμό εμπιστευτικότητα, κάτι το οποίο δεν είναι αυτομάτω κακό. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι και θα ήθελα να εστιάσω λίγο στους κινδύνους. Εγώ είμαι ειδικό ε, του οικονομικού εγκλήματος, ε, το μελετώ εδώ και 25 χρόνια στην Ευρώπη, ανά τον κόσμο και ε, ελευθερλημένες είναι ευε, ευάλωτοι όσον αφορά ακριβώς το ξέβλημα χρήματος και το οικονομικό έγκλημα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε για τα μέρη αυτά. Πολύ εμπόριο που διεξάγεται μεταξύ των διαφόρων μερών και των ιδιοκτητών των ζώων αυτών, το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Αν κάποιος αγοράσει ένα σπίτι στο Βερολίνο, φαίνεται στο υποθυκοφυλακείο, κάποιος το αγόρασε, κάποιος το πούλησε. Αλλά οτιδήποτε γίνεται στους ελεύθερους λιμένες είναι εμπιστευτικό. Ε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την τρίτη και τέταρτη οδηγία έχει πρόσβαση σε αυτές τις ε, πληροφορίες, αλλά έχουν πρόσβαση όπως θα το έκανε παραδείγματος χάρη διεθνής διαφάνεια ή ένας δημοσιογράφος. Όχι, δεν ε, υπάρχει ακριβώς αυτού του είδους η διαφάνεια. Υπάρχουν διαφανεια υπαρχουν βεβαιως οι ε, τελωνιακοί Υπάρχουν διάφορα εμπόδια, ε, υπάρχουν μηχανήματα, ακτινογραφίες κλπ. Αλλά το ερώτημα είναι αν τα γνωρίζουμε όλα. Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε. Έχουν γίνει πολλές μελέτες και δεν ξέρουν πολλοί άνθρωποι την απάντηση στο ερώτημα. Και αυτό δεν είναι απλά ένα σύμπτωμα των ελευθερών λιμένων. Είναι θέμα ξεπλήματος χρήματος. Το ξέπλυμα χρήματος είναι σαν το νερό, όπως κατεβαίνει από το βουνό. Αναζητά πάντα μια... την ευκολότερη εδώ. Τώρα, είτε αυτή είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξής βίζε ή οι ελευθερημένες, ε, θα το βρει και θα το εκμεταλλευτεί. Και σύμφωνα με το ΔΝΤ, αυτή η Παγκόσμια Τράπεζα κτλ. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο που περνάνε μέσα από αυτούς τους κλάδους ετησίως ε, και μιλάω ακριβώς για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών γιατί όλοι μελετούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά δεν μελετάει πολλοί κόσμος τα ζητήματα εμπορίου και υπηρεσιών και γίνεται πολύ ξέπλυμα ε, χρήματος ε, μέσω του εμπορίου και το εμπόριο βεβαίως διεξάγεται στους ελεύθερους λιμένες. Τα χαμένα φορολογικά έσοδα είναι πραγματικά συγκλονιστικά αν μιλάμε δηλαδή για ένα 3 εκατομμύριο δολάρια που περνάει μέσα από το σύστημα, ε, ουσιαστικά αποτεχάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την δίωξη του ξεπλήματος χρήματος. Ίσως να ανοιχνεύουμε το 0,5% του ξεπλήματος που γίνεται αν μιλάμε για ένα 3 εκατομμύριο. Οπότε είναι τεράστιο το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παραπέρα νομοθεσία, λέω εγώ, δεν είναι η λύση. Υπάρχουν πολλοί νόμοι, η ε, πέμπτη ευρωπαϊκή οδηγία είναι φανταστική. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Η επιβολή και η διώξεις είναι το πρόβλημα. Δεν ασκούνται διώξεις για το ξέπλυμα χρήματος, γιατί δεν ε, θα σταματήσουμε ποτέ το φαινόμενο αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μπορούμε να το μετατοπίσουμε σε μια άλλη χώρα, κάπου ή να ασκήσουμε κάποια αποτροπή. Εγώ προτείνω λοιπόν οι νόμοι μας ε, να έχουν χαρακτήρα αποτρεπτικό. Ένας εγκληματίας θα το ξανασκεφτεί εάν γνωρίζει ότι υπάρχουν σοβαρά αποτρεπτικά μέτρα. Επίσης προτείνω να πάμε πέρα από το να ασχολούμαστε με αυτόν ο οποίο διαπράττει το οικονομικό κλίμα, υπάρχουν και αυτοί οι θεματοφύλακε. Τράπεζε, τράπεζες, οι δικηγόροι και οι λογιστές. Συχνά λέω δηλαδή πώ είναι δυνατόν μια, ένα λογιστικό γραφείο να μην προσέξει μια απάτη. Οι δικηγόροι πως λένε, πόσο προσπερνάνε τέτοια ζητήματα. Το ίδιο και με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τώρα έχουν κάνει πολλές προσλήψεις στον τομέα αυτών αλλά κάνουν τίποτα. Εξακολουθούν να βγάζουν δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη. Επενδύουν αρκετά λοιπόν στον τομέα της συμμόρφωσης. Λοιπόν, έχω δει τις ε, πληροφορίες ε, που πηγαίνουν στις υπηρεσίες δίωξης οικονομικού εγκλήματος σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και διαφέρουν ε, κατά πολύ. Έχουν διαφορετικούς πόρους, αλλά δεν επεξεργάζονται επαρκώς ε, τις ύποπτες αυτές συναλλαγέ. Πρέπει να ασχίσουμε πίεση λοιπόν στι τράπεζε, αλλά όπως είπα και στους άλλους ε, φορείς. Οπότε, η νομοθεσία είναι το ένα. Αλλά, για να υπάρξει κάποια ουσιαστική διαφορά, θα πρέπει να υπάρξει ένας αποτρεπτικός χαρακτήρας. Μπορώ να απαντήσω και σε ερωτήσεις, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να χρηματοδοτούν καλύτερα οι μονάδε καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματο σε διάφορες χώρες, είτε στη Μάλτα, είτε στη Λετωνία, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει ομάδα εγγμών που μεταφέρει τα δεδομένα κτλ. Αλλά αυτό γίνεται σπόραδικα. Και βεβαίω ε, υπάρχει και πολιτικό συμφέρον για να μην μεταδίδονται αυτά τα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να γίνεται κέντρικα κάτι τέτοιο, να θέσουμε και να εξαναγκάσουμε τον κόσμο να αναφέρει στις μονάδες αυτές ε, με έναν πιο οργανωμένο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτηθεί και να αλλάξει τελείως η στρατηγική αυτή, γιατί κοιτάμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κανείς δεν κοιτάει το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Επίσης προτείνω η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που πιθανώς αναλάβει το έργο δεν είναι το κατάλληλο θεσμικό όργανο, έχει εποπτικό χαρακτήρα. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει κάποια έρευνα και επιβολή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κίνητρα στις διοκτικές αρχές ε, για να δρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασκούν διώξεις για το οικονομικό έγκλημα. Αυτή είναι η απόψη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Φαβιέν Γκράσερ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Είμαι από την εφημερίδα Λεκοτιδιά του Λουξεμβούργου. Είμαι μεγάλος, αλλά γνωρίζω και εργάζομαι στο Λουξεμβούργο εδώ και 25 χρόνια. Ασχολούμαι με θέματα βρώμικου χρήματος, ασχολήθηκα και με τα LuxLeaks και τα Panama Papers, με θέματα φορολογικά και σε σχετικά με το Freeport έχω αφιερώσει πάρα πολλά άρθρα. Ενδιαφέρθηκα λοιπόν εκ των προτέρων με την υπόθεση των Freeports, είναι μια δομή που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014 και είμαι εδώ χάρη ή εξαιτία της ε, Επιτροπής σας. Με είχε προσκαλέσει η Επιτροπή Πανά για το Freeport, μου τέθηκαν ερωτήσεις, δεν έχω πολλές απαντήσεις δυστυχώς να δώσω. Είναι κάτι το οποίο παραμένει αρκετά μυστικό θα έλεγα. Εν τω μεταξύ ενδιαφέρθηκα περισσότερο στους ε, μετόχους και όχι τόσο τους πελάτες του Freeport και γιατί είναι πιο απλό και υπήρξε μια επίσκεψη στις αρχές του χρόνου ε, βουλευτών της Παλαιάς Επιτροπής Πανά, οι οποίοι ήρθαν εκεί και έθεσαν πάρα πολλές ερωτήσεις στους υπευθύνους του Freeport και ιδιαίτερα σε, για μια επιχείρηση που ασχολείται με τη διαχείριση του χώρου. Την Freeport Management. Οι ερωτήσεις αυτές δεν έλαβαν απαντήσεις τους παρέπεμψαν στην υπηρεσία τελωνίων του Μεγάλου Δουκάτου. Λάβαμε κάποιες απαντήσεις, είναι γενικόλογες κάπως, ε, ε, λένε τα ίδια ότι όλα είναι νόμιμα. Γενικά βάζουν στην άκρη ότι είναι δεοντολογικό, τα είναι ηθικό. Εντάξει, μπορεί και να μην είναι πολύ ηθικό, αλλά είναι νόμιμο. Για την κυβέρνηση λοιπόν του Λουξεμβούργου και για τους υπευθύνου ε, του Freeport αυτή δεν είναι έμποροι. Στην ουσία είναι ένα κομμάτι της επιμελητίας αν θέλετε, της αλυσίδας της επιμελητιακής ε, για να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες της χώρας. Όλα μας λένε ότι είναι διαφανή. Εγώ έχω αμφιβολίες βέβαια για δύο λόγους είμαι σε επαφή με τη διοίκηση του Freeport, μου είπαν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν, απε, δεν απεδείχθησαν αληθή και υπάρχει μια διαρκής αντίφαση από τη μία ανάμεσα στους υπευθύνους της Freeport που λέει ότι εμείς απλά νοικιάζουμε τους χώρους, δεν είμαστε υπευθύνοι για το τι συμβαίνει μέσα σε αυτούς τους χώρους και από την άλλη μας λένε η τελωνιακή υπηρεσία είναι υπεύθυνη και τα ελέγχει όλα αυτά και όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει μια μυστικότητα σε ό,τι έχει σχέση με το Λουξεμβούργο και ιδιαίτερα με το Freeport. Μία από τις ερωτήσεις είναι αν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις στο παρελθόν. Δεν μάθαμε τίποτα. Οι αρχές δεν λένε και πολλά. Πάντως εγώ εργαζόμενος στο θέμα αυτό εδώ και 20 χρόνια ε, περίπου εργάζομαι με ευαίσθητα θέματα, βλέπω την αντίδραση των μετόχων ε, και της κυβέρνησης ε, με απείλησαν γραπτά τηλεφωνικά, με εξύβρισαν υβριστικές επιστολές, απειλητικές επιστολές, με δικαστικούς κλητήρες, με δικηγόρους και πραγματικά κάθε τι που γράφω για το Freeport προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις ε, λοιπόν, γιατί είναι τόσο ευαίσθητοι αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ξέρετε ότι υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στους βουλιέ που είναι οι πραγματικοί ε, αρχικοί ιδιοκτήτες ε, και τους Ρώσους ιδιοκτήτες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ζημίες, οι ζημίες μεγαλώνουν, τα κοντέινερ είναι όλο και λιγότερα ε, υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ευαισθησία γύρω από την υπόθεση αυτή. Τώρα για τον ε, νόμο στο Λουξεμβούργο. Νομίζω ότι είναι από τα λίγα Freeport που ε, υπόκεινται στην οδηγία για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Το Λουξεμβούργο έχει μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις υποδειγματικές για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος αλλά ο κύριος Κάρτο είπε ότι λόγω του μεγέθους του Λουξεμβούργου, λόγω των υποθέσεων με τις οποίες θα καλό είναι να υπάρχουν καλές νομοθετικές διατάξεις, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται, να υπάρχουν έλεγχοι. Ε, το 2010 είχε υπάρξει μια πρώτη έκθεση της Επιτροπής Πανά για τον ε, χρηματοπιστωτικό ε, τομέα που είπε ότι υπήρχαν 16 υπάλληλοι που ασχολούνται με 22.000 πιθανές παραβάσεις το χρόνο. Συνεπώς τίθεται το θέμα. Ναι μεν είναι υποδειγματικό το Freeport σε σχέση με τους νόμους οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία τους, αλλά πραγματικά εφαρμόζονται οι νόμοι αυτοί, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να δω για μένα τον ίδιο Πιστεύουν πολλοί ότι είμαι ειδικό σε θέματα οικονομικών και φορολογίας. Όχι, δεν είναι σωστό. Αυτό το οποίο εγώ κάνω ε, ασχολείται περισσότερο με την καθημερινότητα και με τα τυχαία συμβάντα. Ε, σαν παράδειγμα το πλήσιμο του βρώμικου χρήματος είναι ιστοριούλες με κλέφτες και αστυνόμους. Το πρόβλημα για τον τύπο στο Λουξεμβούργο είναι ότι πολύ συχνά υπάρχουν κλέφτες αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πάρα πολύ συχνά αστυνόμοι οι οποίοι να τους κυνηγούν. Τα πράγματα εξελίσσονται από μόνα τους και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί και με το Freeport, θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες πληροφορίες, τις οποίες δυστυχώς λόγω της μυστικότητας που διέπει τη λειτουργία του δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής, όπως πάντα. Θα υπάρξει χρόνος για ένα λεπτού ερώτηση και τέσσερα λεπτά απάντησης. Εισηγητές, Νίντε Μάια. Ευχαριστώ, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ερώτηση για τον κύριο Καρ και πρώτα. για τα θέματα εξηγήσατε την περιπλοκότητα της αντιμετώπισης ε, του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Μπορείτε να εξηγήσετε τι έχει συμβεί. Υπάρχει βελτίωση της νομοθεσίας, περισσότερη διεθνή συνεργασία. Έχουμε αυτοματοποιημένες ανταλλαγές ε, ε, πληροφοριών λογαριασμών των κυρίων. Έχουμε επίσης πληροφορίες για τους μετόχους και κυρίους των εταιριών. Για σας, ποιες είναι οι σημαντικότερες ελλείψεις διότι βεβαίω το σύστημα, όπως μια λυσίδα, θα είναι τόσο ισχυρό όσο, όσο είναι το, το ε, πιο αδύναμο σημείο του. Η EBA, είπατε, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, δεν είναι ε, ο καλύτερο οργανισμό για να παίξει σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση του, της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Συμφωνώ μαζί σας, ήμουν και εγώ κεντρικός τραπεζίτης. Αντιλαμβάνομαι ότι η εποπτεία είναι προληπτική, ενώ το, η αντιμετώπιση του είναι κάτι διαφορετικό. Πρώτα όμως χρειάζεται διερεύνηση ε, υποθέσεων. Μετά όμως χρειάζεται και κάποιος ο οποίος θα εξετάζει την ποιότητα των συστημάτων μέσα στις τράπεζες σχετικά με τη συμμόρφωση των διαδικασιών τους με το δίκαιο. Ποιο είναι ο πλέον κατάλληλος για να αναλάβει αυτή τη ε, δράση. Ευχαριστώ κύριε Κάρεσης. Όντω έχουν γίνει μεγάλα βήματα σε όλου του τομεί που εξηγήσατε σε ό,τι αφορά την διαφάνεια UBO, δηλαδή ο ε, απότατος ε, δικαιούχος, ο τελικός δικαιούχο, το ξεκαθάρισμα διαφόρων ειδών εταιριών να μην παραμένουν ε, καταθέσεις σε τράπεζες που να είναι άγνωστες, να μπει διαφάνεια δηλαδή ε, στα τραπεζικά συστήματα βεβαίως και η ε, κοινοποίηση των ε, λεπτομεριών αυτών. Εκεί όπου μπορεί να γίνει επένδυση και χρημάτων και ε, χρόνου είναι η ανάλυση των δεδομένων. Διότι μιλούμε για ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Τεράστια, τεράστια, τεράστιου όγκους δεδομένων. Βέβαια έχουμε το πλεονέκτημα σήμερα ότι έχουμε στην διάθεσή μα πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούν να αναλύσουν τα δεδομένα αυτά. Όμω πρόκειται για δουλειά ειδικών προσόντων. Δυστυχώ οι τράπεζε ε, έχουν κάποια σύγκρουση και οι σχετικές μονάδες δεν είναι επαρκώς επανδρομένες ή δεν έχουν επαρκείς πόρους. και τα δύο. Δεν έχω ακρίβή στατιστικές, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες συναλλαγών που ε, καταγράφονται κάθε χρόνο και δεν έχουμε επαρκείς πόρους για να τις συζητήσουμε όλες. Εννοώ τις ύποπτες. Και οι τράπεζε παίζουν ένα κάπω διπλό ρόλο. Δηλαδή βασίζονται σε αυτό για να μην τι κοινοποιούν όλε. Εκεί όπου μπορούσε να γίνει μια επένδυση σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι να εξασφαλιστούν τα αναγκαία προσόντα από το προσωπικό των ε, ε, μονάδων που θα εξετάζουν τα θέματα αυτά. Αυτή είναι η πρώτη μου σύσταση τώρα για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Βεβαίω χρειάζεται εποπτεία. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή εξετάζει μια πτυχή, δεν εξετάζει το εμπόριο με overpricing και underpricing της αξίας, ανατίμηση, υποτίμηση της αξίας, ή επενδύσεις σε μετοχές, ή λήψη δανείων από hedge fund, ή συλλογικές έργων τέχνης και όλα τα λοιπά. Όλα αυτά ξεφεύγουν από το ραντάρ. Η EBA μπορεί λοιπόν να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εποπτεία και το να εξετάζει τι συμβαίνει στον χρηματοπιστωτικό κόσμο, αλλά το ξέπλυμα ε, βρώμικου χρήματο είναι σαν το νερό. Πάει και βρίσκει το ε, πιο αδύναμο κρίκο και τον διαλύει και, και περνάει μέσα, από μέσα. Η ποιότητα λοιπόν της διερεύνησης χρειάζεται συντονισμό σε ένα συλλογικό όργανο. Οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, έχουν ένα κεντρικό ε, σύστημα anti-money laundering, το οποίο εξετάσει όλο το φάσμα και το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και η Ευρώπη. Νίτερ Μάιερ, διευκρινιστική. Εσείς εννοείτε να συγχωνευτούν αυτές οι δύο λειτουργίες. Το ένα είναι καταστολή, το άλλο είναι εποπτεία. Έχουν μια διαφορά, αλλά χρειάζεται να υπάρχει ένα συσχετισμός μεταξύ τους. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση. Αυτό με απασχολεί γιατί είναι και ο χαρακτήρα μου έτσι. Ή, μπορεί ίσω τραπέζε να το κάνουν καλύτερα. Ή, ή τα Freeport. Όποιο χρειάζεται δηλαδή να περνά καλύτερη ποιότητα δεδομένων. Και τα δεδομένα αυτά να αναλύονται έτσι ώστε να μπορούν να οδηγούν και σε διώξει. Ευχαριστώ. Σοσιαλδημοκράτε. Κόφουτ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και το πανελ για τι ειδικέ οικονομικέ ζώνε όλα τα δεδομένα που μας δώσατε πραγματικά δεν ξέρω αν δικαιολογούν ότι υπάρχει κάποια οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις ειδικέ οικονομικές ε, ζώνες και ε, το είπαμε και στην Επιτροπή μας, ε, στην προηγούμενη Επιτροπή το είδαμε αυτό το θέμα με την κατάσταση που έχουν στην Πορτοκαλία όπου δεν βλέπουμε κάποια οικονομική ανάπτυξη εκεί παρά το ότι αυτό υποτίθεται ότι πρόκειται. Λοιπόν, ε, πολύ ενισχυτικό αυτό. Ε, στην διαφάνεια εδώ πέρα μιλάτε για φορολογικά κίνητρα, το οποίο σημαίνει τα πάντα έτσι. Ε, κίνητρα όσον αφορά τον εταιρικό φόρο ή οτιδήποτε άλλο. Για τους ελεύθερους λιμένες. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κάποιο όριο στο τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Ε, πόσο καιρό μπορούν να λειτουργούν αυτά τα ελεύθερα λιμάνια. Γνωρίζουμε, παραδείγματο χάρη, ότι εκεί πέρα φυλάσσονται έργα τέχνη, κοσμήματα, χρυσό, ε, πολλά και διάφορα πράγματα. Πού καταγράφεται αυτό και πόσο καιρό μπορούν να λειτουργούν και πόσες φορές μπορούν να απολυθούν και να αγοραστούν κάποια πράγματα και αν υπάρχει κάποιο όριο. Γιατί βλέπουμε ένα παράλληλο σύστημα το οποίο όπως γνωρίζουμε στην Επιτροπή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Μετά κύριε Κάρ, ισχύει το ότι δεν υπάρχει επιβολή και δίωξη και ανείχνευση υποθέτω έτσι. Γιατί είπατε και ο ίδιος τους αριθμούς ότι πρακτικά δεν υπάρχει κίνδυνος ε, στο ξέπλυμα χρήματος. Αναφέρατε λοιπόν τις μονάδες ε, οικονομικού εγκλήματος. Χρειάζεται, θα λέγατε, κάποιο είδους ε, FBI στην Ευρώπη για τα οικονομικά εγκλήματα, γιατί έχετε δίκιο. Βεβαίω έχουμε σκάνδαλα στις τράπεζες. Μπορούν να έχουν στα χαρτιά την τέλεια πολιτική συμμόρφωση, αλλά αν δεν την εφαρμόζουν δεν έχει καμία σημασία. Χρειάζονται λοιπόν επιτόπιοι έλεγχοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των ελεύθερων λιμένων και των λοιπόν, για να δούμε αν πραγματικά ακολουθούν την νομοθεσία, γιατί μέχρι στιγμής ε, η πολιτική μας αποτυγχάνει και εμπιστευόμαστε ε, την αυτορύθμιση υπερβολικά και αποτυγχάνουν ε, τα χρηματοπιστωτικά θέματα. Μήπω λοιπόν χρειάζεται να πηγαίνει κάποιο επί τόπου για επιθεωρήσει και για την Κομισιόν, ναι, ξέρω βεβαίω ε, τα όρια τη εθνική ε, δικαιοδοσία, αλλά για να έχουμε μια πραγματική κοινή αγορά ε, δεν είναι πρόβλημα το να μην έχουμε ελέγχου όταν η νομοθεσία που κάνουμε δεν εφαρμόζεται και δεν διώκονται οι παρανόμες δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν την Κομισιόν, τον κύριο Κέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για να προσπαθήσω να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις. Το ένα αφορά το καθιστώς των ελεύθερων ζωνών. Γιατί στον Ευρωπαϊκό Τελωνιακό Κώδικα έτσι ορίζονται στις ελεύθερες ζώνες. Δεν υπάρχει χρονικό όριο για το πόσο θα παραμείνουν εκεί τα αγαθά. Υπήρξε πλήρη αναδιατύπωση τη σχετική νομοθεσίας στον τελωνιακό κώδικα και εκεί πέρα θα δείτε ότι η έννοια της ελεύθερη ζώνης πηγαίνει μαζί με τις ε, τελωνιακές αποθήκες ως ε, κάποιο είδου αποθήκευση. Δηλαδή έρχονται στην ελεύθερη ζώνη τα αγαθά, μπορούν να παραμείνουν εκεί, αλλά εάν βγουν ε, τότε ε, αντιμετωπίζονται ως εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρομοίως, η διαδικασία κατά κανόνα είναι ότι οι διατάξει περί ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης ακολουθούν, θα έλεγα, τις ε, διατάξεις περί τελωνίων, αλλά στην περίπτωση του ΦΠΑ υπάρχει διαβούλευση της Επιτροπής ε, ΦΠΑ και πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Για το θέμα δε των επιθεωρήσεων, όσο έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και από τη σκοπιά που τα βλέπω εγώ, την τελωνιακή, υπάρχουν δύο τομείς μπορούμε να δούμε. Το ένα είναι η διαδικασία που κάνει η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, αλλά αυτό είναι παραδοσιακή πολιτική των ίδιων πόρων. Και βεβαίως το δεύτερο είναι οι έρευνες του Όλαφ που αφορούν συγκεκριμένες απάτε. αλλά πέρα από αυτά δεν γνωρίζω κάποιες αρμοδιότητες που έχουμε για να δούμε τις ε, διαδικασίες, γιατί όπως ε, το βλέπω αυτή τη στιγμή η νομοθεσία γίνεται σεβαστή όσον αφορά τις ε, διατάξεις που ισχύουν την υποχρέωση να είναι κλειστή η ελεύθερη ζώνη και να υπάρχει τελωνιακή εποπτεία. Συμφωνώ μαζί σας. Ακριβώ η ανείχνευση είναι εδώ πέρα θεμελιός λίθος της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και είναι κάτι το περίπλοκο σήμερα γιατί απαιτεί βαθύτατη ανάλυση πολλών πληροφοριών και είναι πραγματικά ευθύνη των διαφόρων διαμεσολαβητών που πρέπει να την πούμε στον Ιά. Φέρω δύο παραδείγματα. Πώς μπορεί στην Εσονία και στην Λετωνία να υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια ε, ρωσικών και ουκρανικών κεφαλαίων να περάσουν από ένα υποκατάστημα. Πώς μπορεί να συμβεί δηλαδή κάτι τέτοιο και να μην το ανοιχνεύσει το σύστημα. Πώς μπορεί να μην το δει η κεντρική τράπεζα και να χτυπήσουν καμπανάκια. Οπότε η ανείχνευση εκεί στην πρώτη γραμμή είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα αν απαιτείται ένα FBI στην Ευρώπη για τα οικονομικά εγκλήματα δεν ξέρω, κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε με το status quo. Και αν ε, δοθεί προτεραιότητα σε περισσότερους πόρους, στις τράπεζες ή στους ενδιάμεσους ε, ή και στους δικούς μας ερευνητές, νομίζω θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες δεν είναι εδώ. Βέρνερ Λάγκεν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την πείρα της ε, Εξεταστικής Επιτροπής ε, στο Λουξεμβούργο θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Είχαμε πάει επί τόπου, είδαμε το παράδειγμα του Ελεύθερου Λιμένα, ο οποίος είναι αποκλεισμένος, ε, ασφαλισμένος, δεν είναι δυνατή πρόσβαση στον καθένα έχει σχετικά υψηλά νίκια, 11 έως 20 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για τους χώρους αποθήκευσης. Είδαμε αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος Κομισιόν ότι υπάρχουν εκεί τελωνιακές αρχές, αλλά όλος αυτός ο ελεύθερος λιμένας μπορεί να είναι μια χαρά νόμιμος, αλλά εποπτεύεται από τρεις τελωνιακούς και υπήρχε ένα τεράστιο σκάνερ που μας το παρουσίασαν ως μεγάλη επιτυχία με το οποίο ανοίχνευαν μεγάλα πακέτα δύο επί 2 μέτρα. Αλλά ε, στην ουσία δεν ξέρει κανείς ε, το τι συμβαίνει εκεί μέσα και το τι αποθηκεύεται. Είναι κάτι παρόμοιο με τις θηρίδες ε, παλιά όπου είχε ένα κλειδί ο ιδιοκτήτης ε, και τράπεζα, αλλά κανεί δεν έλεγχε το τι ήταν μέσα στην θηρίδα. Και εδώ πέρα υποθέτουμε ότι επειδή υπάρχει η παρουσία των τελωνίων υπάρχει σοβαρότερο έλεγχος, παρά το ότι είναι πολύ μεγαλύτερε οι διαστάσεις ε, σε σχέση με τις ε, τραπεζικές θηρίδε. Οπότε οι προτάσεις που έγιναν να υπάρξει κάποιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ίσως είναι σωστό να μην είναι μόνο οι εθνικές αρχές στο Λουξεμβούργο, να το υπενθυμίσω, στα Panama Papers, είχαμε 403 ε, περιπτώσεις, ε, εκ των οποίων οι 300 αφορούσαν δικηγόρους, ε, φοροτεχνικούς κτλ. Υπήρχαν λοιπόν 13 καταδίκες. Στη δε φορολογική αρχή υπήρξε, υπήρξε μόνο μία καταδίκη. Λοιπόν, αν τα αφήσουμε στα κράτη-μέλη, θα ακολουθήσουν όλοι το μοντέλο αυτό του ελεύθερου λιμένα του Λουξεμβούργου. Γιατί βεβαίως δεν μπορεί κανείς να τους προσάψει τίποτα. Σου λέει είναι το τελωνίο στην πόρτα και άρα όλα ελέγχονται. Οπότε θα έπρεπε ε, να υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, το θεωρώ σωστό. Ακούσαμε και την άποψη ειδικών, αλλά θα ήθελα να την Πράγματι υπάρχουν τρεις ε, τελωνοφύλακες. Εξετάζουν από πουρα μέχρι ε, ε, καλλιτεχνήματα, κοσμήματα, ακόμα και πληροφοριακά δεδομένα. Τι, το θέμα τι γίνονται οι πληροφορίες αυτές. Πρόκειται για τελωνιακούς. Δεν είναι ούτε διδάκτορες της ιστορίας, ε, της τέχνης, ούτε άλλο σχετικό πράγμα. Και μια διευκρίνηση που ίσως απαντά στην ερώτησή σας. Μπορεί να αποθηκεύσει κανείς επαόριστον, μπορεί όμως και να πωλεί και να αγοράζει στο εσωτερικό μεταξύ διαφόρων φορέων. Γίνεται μια δήλωση, γίνεται μια τελωνιακή διασάφηση, μπορούν όμως τα πράγματα αυτά να παραμείνουν επάπειρον, επαόριστον ας πούμε έτσι, μέσα στο Freeport. Κάτι άλλο που πρόσεξα, υπάρχει μια διαδοχική σειρά επιχειρήσεων, εταιριών που ελέγχουν το Freeport. Όταν μιλεί κανείς για δεδομένο, φτάνει αμέσω σε χιλιάδες ε, σελίδες δεδομένων που περιγράφουν ποιος κάνει τι κτλ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η έλεγχη υπάρχει ο ελεύθερος λιμένας, το Freeport. Γίνονται τακτικά επισκέψεις διεθνών φορέων, που συγχαίρουν για την ασφάλεια, είναι πραγματικό Fort Knox κλπ. Και υπάρχει και διαφάνεια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνίων και μάλιστα έχει γραφτεί και σε μια από τις απαντήσεις η αντιπροσωπεία των γαλλικών τελωνίων ήρθε στο Freeport για να τον συγχαρεί για την διαφάνειά του. Υπήρξε προφορία αυτή. Έκανα επαλήθευση, ποτέ δεν έφτασε αντιπροσωπεία των γαλλικών τελωνίων εκεί. Ποιο μπορεί να, ελέγξει λοιπόν οι λουξεμβουρικέ αρχές. Δηλαδή το κάνουν. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο που να μιλεί για τον ε, έλεγχο. Ο κύριος Μπουργέ έχει προσκληθεί εδώ αξιωματούχος των γαλλικών τελωνίων. Γνωρίζω ότι ήρθαν κάποιοι από αυτούς, ήρθαν και είπαν ότι είναι εντάξει. Και τώρα ισχυρίζεται το λουξεμβουργικό Freeport ότι έχει την σφραγίδα ποιότητα των γαλλικών τελωνίων. Ψευδέ. Ήρθα σε επαφή με τα γαλλικά τελωνία και η προφορία αυτή είναι ψευδή. Υπάρχει και κάτι άλλο. Στις ανταλλαγές απόψεων που έχω κάνει μαζί του, μου είπαν ότι οι άνθρωποι τη Εξεταστική Επιτροπής Πανά δέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος για το Freeport του Λουξεμβούργου και ότι όλα ήταν καλά. Δεν ξέρω ποιος από τη δική σας επιτροπή Πανά πήγε και τους είδε και είπε αυτά τα πράγματα. Γίνεται πολλή επικοινωνία γύρω από το Freeport. Φαίνεται πως προσκαλούνται ε, λουξεμβουρικές εφημερίδες, μας δείχνουν ε, αποκαταστάσεις πινάκων κλπ. Να πω κάτι και για τους άλλους μετόχους, η Βουβιέ για παράδειγμα, ο οποίος ε, συντάσσει και μια ε, δικαστική επιθεώρηση εδώ και πολλά χρόνια και για το θέμα των πινάκων και υπάρχει και μία διαφορά ε, της τάξης των 400 εκατομμυρίων. Υπάρχει άλλος ε, μέτοχος, Λιβιέτο Τομά, γαλλικής που κατηγορείται τώρα και διώκεται για κλοπή πινάκων του Πικάσο. Υπάρχει και ένα τρίτος που λέγεται Περετή και ο οποίος εμφανίζεται συχνά σε έγγραφα, σε ντοκιμαντέρ γαλλικά ο οποίος συνδέεται με κορσικανικές ε, συμμορίες. Ε, το γεγονός είναι ότι ο κύριος αυτός ηγείται κύκλου καζίνο στο Παρίσι που έκλεισε το 2008-2009 μετά παρέμβαση των αρχών και τον οποίον, το όνομα του οποίου δηλαδή, βρίσκει κανείς ξανά και ξανά σε άρθρα στη Γαλλία σχετικά με, οργανο, ε, με ε, οργανωμένου κλίματος στην Γαλλία, εμφανίζεται και σε έργα για, τη... για σε... σε μάλλον για την ε, μαφία του ποδοσφαίρου και το καθεξής. Αυτά είναι τα ονόματα των μετόχων του Freeport Λουξεμβούργου. Πρόεδρος. Λάνγκεν. Μετά από την επίσκεψη έγινε και μια συζήτηση με τον ε, τύπο που είχε οργανώσει το ίδιο το Freeport. Δεν ήμουν δυστυχώς παρόν και δεν μπορώ να διαβεβαιώσω ότι υπήρξε σχετική ενέργεια. Απάντηση του κ. Κρασέρ χωρίς μικρόφωνο. Όπως είπαν πολλές, πολλοί βουλευτές ότι είχε χτυπηθεί άσχημα εν πάση περιπτώσει κατά τη διάρκεια της ε, ε, συνέντευξης τύπου. Όλοι έλεγαν ότι όλα είναι διαφανή, ότι ο έλεγχος είναι πλήρης, αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν ξέρω το τι μπαίνει μέσα στο Freeport και τι γίνεται. Οπότε στην ουσία υπάρχει μια μετάθεση της ευθύνης ανάμεσα τα τελωνία, στο Υπουργείο και στη διαχείριση της Freeport. Ε, νομίζω ότι η εταιρεία η οποία ελέγχει είναι μια εταιρεία η οποία αποτελείται από δεκάδες άλλες εταιρείες, χιλιάδες καταστατικά από δεκάδες χώρες. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Αυτές ε, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ουσία, δεν έχουν κανένα υπάλληλο, απλά είναι επιχειρήσεις ε, ταχυδρομικά κοιτία. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις ότι δεν είχε υπάρξει σε σχέση με το θέμα αυτό επίσημη δήλωση της Επιτροπής Πανά. Να διευκρινίσω κάτι εδώ, λέει ο κύριος Πιατσάρντι. σχετικά με τις οικονομικές, τις ειδικέ οικονομικές ζώνες. Δεν είναι κάτι το οποίο μας το οποίο στηρίζουμε ε, με συγκεκριμένο τρόπο. Όχι. Εγώ παρουσίασα μία μελέτη ε, δραστηριότητας 20 ετών και στην έρευνα αυτή υπάρχουν ορισμένες, ορισμένοι δείκτες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι και για τις δικές σας χώρες πώς κάποιες ειδικέ τέτοιες οικονομικού ενδιαφέροντος περιοχές μπορούν να λειτουργήσουν. Μια τέτοια μελέτη ε, χρηματοδοτήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, όχι από μας. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω θα πρέπει να είμαστε σχετικά πραγματιστές σε επίπεδο γεωγραφικό. Τι εννοώ. Όταν ψάχνουμε μία Ήπειρο σαν την Αφρική και μιλάμε για τα σημεία ανάπτυξης, μιλάμε για εμπορικούς ε, μεταφορικούς διαδρόμους, όπως επίσης και για λιμενικές εγκαταστάσεις και οικονομικού ενδιαφέροντος ε, ε, ειδικού τύπου εγκαταστάσεις. Είναι μια πραγματικότητα για χώρες όπως η Αιθιοπία. Αυτό το οποίο έχει όμως σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο διοικούνται όλα αυτά, όλες αυτές οι μονάδες. Και ακριβώς υπάρχουν δείκτες οι οποίοι δείχνουν την αποτελεσματικότητα των μονάδων διαχείρισης. Εμείς δεν κάνουμε κανένα παζάρι ανάμεσα στην ανάπτυξη από τη μία με τους όρους διακυβέρνησης και διοίκησης από την άλλη. η κυρία Ρέγνερ. Είχα πάει με την αντιπροσωπεία στο Freeport Λουξεμβούργου και αισθάνθηκα λίγο σαν σε ταινία του James Bond, ήταν πραγματικά συναρπαστικό πώ ε, γίνεται να μπει κανεί μέσα και λυπούμε που δεν είναι παρόν κανείς εκπρόσωπος είτε των Λουξεμβουργικών Αρχών είτε του Freeport, γιατί βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα που ε, στρέφονται γύρω από τέτοια θέματα που θα μπορούσαν να φωτίσουν. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι το τι βρίσκεται μέσα το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες του Freeport. Και ότι στην ουσία πρόκειται για μια μαύρη τρύπα. Δεν υπάρχει πολύ διαφάνεια. Ερώτηση λοιπόν. Και σας παρακαλώ Όπω βρίσκεστε εδώ υπό τις διαφορετικές ιδιότητές σας, να μας φωτίσετε περισσότερο. Έχετε ιδέα τι κρύβεται εκεί. Μας είπατε ότι σας έδειξαν ε, την αποκατάσταση ενός πίνακα. Και αυτή οι Πικάσο δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα μουσείο ή έστω ε, στην ε, βίλα κάποιου πλουσίου προσώπου. Τι νόημα έχει να κρύβονται μέσα σε ένα freeport τέτοια ε, καλλιτεχνήματα. Και τέλος, το ουσιώδες δίκαιο, αυτή η πέμπτη οδηγία για, κατά της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων, αρκεί, διότι μιλούμε για υψηλής αξίας ε, υποθέσεις. Ο κύριος Λάγκεν άλλωστε το έδειξε προηγουμένως, μιλούμε και για τους διαμεσολαβητές. Τα όσα είδαμε εκεί ήταν, ιδιαίτερα, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι πρόκειτο για ε, εταιρείε γραμματοκιβωτίου. Αυτές κάνουν τις ε, επαφές μεταξύ των ιδιοκτητών και των τελωνιακών αρχών. Ουδής γνώριζε τι είδους αντικείμενα βρίσκονται αποθηκευμένα εκεί. Αισθανόμουν σαν εκείνα τα τρία πυθικάκια που λένε μην μιλάς, μην ακούς και μην βλέπεις. Ε, ότι κάπως σε τέτοιες εντολές υπακούν δηλαδή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε περισσότερα στη βάση των ε, υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κύριε ε, Γκρασέρ. Για να ολοκληρώσω, γιατί υπάρχουν παρόμοια ερωτήματα από την επίσκεψη και τα άρθρα για το Freeport. Το Freeport οι πόρτες του Freeport έχουν κλείσει πλέον ερμητικά. Τώρα, γιατί ο κόσμος αποθηκεύει ε, καλλιτεχνήματα σε τόπους όπως τα φρυπόρτες έχουν κάτι να κρύψουν. Πρόκειται όμως και για μια, ε, να μια, μια τροπή που έχει πάρει η αγορά έργων τέχνης που γίνεται πλέον ηλική επένδυση. Κανονικά ναι, τα έργα θα έπρεπε να είναι στα μουσεία. Κάποια φορά θέλουν να τα κάνουν γιατί είναι και ιδιοκτησία τραπεζών και αυτά θέλουν να τα δείξουν για να κάνουν και διαφήμιση. Νομίζω όμω ότι τα Freeport είναι και πραγματικά ο ιδανικό τόπος για να αποφύγουν την προσοχή των φορολογικών αρχών. Κάτι άλλο που υπάρχει σε σχέση με τα Freeport, μιλήσαμε για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, φορολογικών αρχών δηλαδή, αλλά τα Freeport ξεφεύγουν ακόμα από την υποχρέωση αυτή διαφάνειας. Ας πούμε ένας Ισπανός μπορεί να αποθηκεύσει κάτι στο Freeport του Λουξεμβούργου. Το γνωρίζουν οι Ισπανικές φορολογικές αρχές. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό για αυτή την ώρα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά που πρέπει να ρυθμιστούν ακόμη σχετικά. Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Η Φιλελεύθερη, ο κύριος κρίντς Σας ευχαριστώ πολύ το ότι, ότι έχουμε μπροστά μας υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος δεν είναι και τίποτα το νέο, αλλά μου σηκώνουν τα μαλλιά όταν ακούω τις τάξεις μεγέθους. Μιλούμε για παροχές ε, υπηρεσιών τάξεως δισεκατομμυρίων ή και τρισεκατομμυρίων. Ερωτώ, γνωρίζομαι ότι οι ελεύθεροι λιμένες χρησιμοποιούνται και για παράνομες ή ύποπτες δραστηριότητες. Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν με τα τυχερά παιχνίδια κάποιες δικαιοδοσίες που αντιλαμβάνονται ότι έχουν σχέση με εγκληματικέ ενέργειε, γιατί δεν τα απαγορεύουμε. Γιατί δεν απαγορεύουμε, τουλάχιστον στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδρυση τέτοιων Freeport. Καταλαβαίνω ότι ίσω στην Αιθιοπία να είναι αναγκασμένοι να το, να το κάνουν αλλά γιατί δεν το υποχρεώνουμε. Και να κάνουμε και κάτι ακόμα. Δεύτερο, για να αποφευθεί ο κίνδυνος συμπεγνία μεταξύ φορολογικών αρχών, ακόμα και μελών κυβερνήσεων και τέτοιων επιχειρήσεων, είναι πολύ μεγάλος. Το είδαμε αυτό και στην ε, περίπτωση ε, κυβερνητικού στελέχους του Λουξεμβούργου. Οι ποινέ για τους ιδρυτές τέτοιων Freeport θα πρέπει να αυξηθούν πολύ σημαντικά σε περίπτωση που αποκαλυφθούν ε, εγκληματικές δραστηριότητες. Ας ξεκινήσουμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Πρώτο λοιπόν. Δεύτερο, κατανοώ ότι είπε ο Charles Carr ότι χρειαζόμαστε όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες μια ισχυρή ευρωπαϊκή αρχή η οποία θα αναλάβει τον αγώνα κατά των ε, δραστηριοτήτων αυτών. Είναι ωστόσο χρονοβόρο, χρονοβόρα η διαδικασία δημιουργίας τέτοιας αρχής, διότι χρειάζεται να περάσει από πολλές φάσεις διαδικασίας, να εγκριθεί τελικώς και από τα τρία θεσμικά όργανα και ούτω καθεξής. Για την παρούσα κοινοβουλευτική θητεία που λύγει τον, την επόμενη άνοιξη δεν θα προλάβουμε. Γι' αυτό ρωτώ, έχει νόημα τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα να ανατεθεί το καθήκον αυτό στην Ευρωπαϊκή ε, τραπεζική αρχή, ώστε τουλάχιστον να βάλουμε το πόδι στην πόρτα πριν να κλείσει. Και το τρίτο, πώς είναι δυνατό οι Financial Intelligence Units στην Ευρώπη, στις διάφορες χώρες, να είναι τόσο ασθενώς στελεχωμένες και να μην μπορούν να εργαστούν. Δεν είναι δυνατόν εκεί να διορθωθεί η κατάσταση ταχαίως. Ευχαριστούμε πολύ, λέει πρόεδρος. Ποιος θέλει τον λόγο, κύριο Σκάρ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσει ξεκινώντας από την τρίτη. Ε, οι μονάδες ε, οικονομικού εγκλήματο, ε, εξαρτώνται από τους προπολισμούς των χωρών. Οπότε στελεχώνονται εσωτερικά από την κάθε χώρα, έχουν ποικίλου προπολισμού ο προπολογισμό του κυμαίνεται και εξαρτάται από την κάθε χώρα βεβαίω το πόσο αποτελεσματική είναι. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά αν έχουμε μια μικρότερη χώρα με λιγότερους πόρους, από την οποία περνάνε πολλά λεφτά, είτε μιλάμε για βαλτικές χώρες, είτε για νησιωτικές χώρες, ε, δεν έχουν αρκετά χρήματα για να ερευνήσουν αυτά τα ζητήματα. Οπότε ίσως ε, θα μπορούσε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρεθεί ένας τρόπος ε, χρηματοδότησης έτσι ώστε να βρεθούν κάποιοι ε, ικανοί άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα και να υπάρξει και μια κατάρτιση. Βεβαίω για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει το status δεν μπορεί η Εστονία, Λετωνία, Μάλτα και ε, συνεχώς να περιμένουμε το επόμενο πρόβλημα και να λέμε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει εποπτικό ρόλο. Οτιδήποτε κάνει τη διαφορά είναι σημαντικό. Υπάρχουν διάφορες συνδομές αλλά δεν αγγίζουν το ζήτημα και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες απαιτήσει από τους ενδιάμεσους ε, τράπεζες, ε, λογιστές, ε, οποιοδήποτε είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και να επανέλθω και στο θέμα της τέχνης. Εκεί πέρα μιλάμε για μια αγορά τέλεια για να μετακινηθούν τα χρήματα. Και έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στην ε, τέχνη και οι ελεύθεροι λιμένες ε, την αποθηκεύουν εκεί, εντάξει γιατί είναι, υπάρχουν την ασφάλεια και αυτό είναι κάτι το θεμητό βεβαίω. Αλλά είναι και ένα μέρος όπου αγοράζονται και πολλούνται γρήγορα τα πράγματα ε, σε τιμές που κανείς ε, δεν αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, αν μιλάμε για έναν πίνακα, έναν πικάσο, πόσο αξίζει. Δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε το ποσό. Και οι αρχές ε, που τα εξετάζουν δύσκολα μπορούν να έχουν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται. Αν κάποιος από το Hong Kong αγοράζει ε, έναν Πικάσο από την Αγγόλα, χρησιμοποιεί τον ελεύθερο λιμένα. Και λοιπόν απαιτούνται εδώ πέρα επιτόπιοι έλεγχοι και μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτές τις συναλλαγές. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Κοιτάξτε, είναι μία μη οικονομική υπηρεσία. Μιλάμε για επιμελητιακές υπηρεσίες, συνεπώς διαφεύγουν πλήρως των ε, παραδοσιακών οικονομικών ελέγχων ε, που ασχολούνται με ε, οικονομικά ιδρύματα, τράπεζες, ασφάλειες κτλ. Μιλάμε για την επιμελητία, τα logistics και σχετικά με την αποθήκευση έργων τέχνης στην Γενέβη, στην αντίστοιχη επιχείρηση υπήρχαν εκατομμύρια έργα τα οποία έχουν μοιραστεί τώρα ανάμεσα στο Σιγκαπούρη, το, το Λουξεμβούργο κτλ. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις να κάνω. Σχετικά με το Freeport, θα μπορούσατε εσείς στα πλαίσια των ερευνών σας να μας πείτε κύριε Γκρέσλερ αν υπάρχει μια υπηρεσία στο Λουξεμβούργο η οποία να είναι υπεύθυνη για να βρίσκει πελάτες για το Freeport και η οποία να έχει έδρα και σε άλλες χώρες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Υπάρχει λοιπόν κάτι τέτοιο, μια τέτοια οργάνωση. Και για τον κύριο Κάρ, σχετικά με την καταπολέμηση ε, του βρώμικου χρήματος. Να πω ότι τα πιστοτικά ιδρύματα στην Ευρώπη ε, έχουν ε, ευαισθητοποιηθεί και νιώθουν υπεύθυνοι για τέτοια προβλήματα. Τις τελευταίες μέρες, σαν παράδειγμα, πήραμε εμείς κάποιες προτάσεις για αποτρεπτικά, αν θέλετε, μέτρα και υπήρξαν τράπεζες οι οποίες καταδικάστηκαν σε πρόστιμα 750 εκατομμυρίων και στη Δανία και στην Λετονία έκλεισαν τράπεζες, η τράπεζα της Μαδρίτης, η τράπεζα της Ανδόρας. Συνεπώς λοιπόν στο πιστοτικό σύστημα υπάρχει ε, πράγματι ένας φόβος ε, που λειτουργεί αποτρεπτικά. Ε, εγώ δεν ξέρω αν γίνεται το ίδιο με τις μεγάλες επιχειρήσεις συμβούλων, δικηγόρων και τα λοιπά, τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες γιατί και αυτές με χρήμα ασχολούνται, έτσι ώστε να ελέγχεται το χρήμα αυτό και να μην προσφέρεται για εύκολο ε, ξέπλυμα. Κοιτάξτε, για το θέμα της προώθησης των δραστηριοτήτων του Freeport ε, για τις επιχειρήσεις ετικέτες υπάρχει μία που λέγεται Luxembourg Management Company ο Ρόλος της είναι να βρίσκει πελάτες. Ε, τώρα για την τέχνη και την ε, αγορά της τέχνης έχουμε να κάνουμε με μια αγορά η οποία είναι πολύ ελεύθερη και δεν είναι ελεγχόμενη. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί έμποροι που πηγαίνουν σε μεγάλες εκθέσεις, συνεργάζονται με γκαλερίστες στην Ευρώπη κτλ αλλά ξέρουμε ότι ε, έχουν προβλήματα και από τις εννέα επιχειρήσεις οι οποίες νοικιάζουν οι τρεις ε, ανήκουν στον Ιμπουβιέ και ασχολούνται με θέματα αποκατάστασης ε, έργων τέχνης κτλ. Πάντα logistics δηλαδή επιμελητία. Όλα αυτά γίνονται με πολύ διακριτικό τρόπο. Ε, δεν υπάρχουν φυσικά διαφημίσεις στην τηλεόραση σε εφημερίδες για τις επιχειρήσεις αυτές. Σχετικά με την ερώτησή σας για το τι άλλο μπορεί να γίνει σε σχέση ε, με τον φόβο ο οποίος θα πρέπει να, να χαρακτηρίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Κοιτάξτε, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ ψηλά, δις δολάρια έχουν, ε, μικρές τράπεζες κλείνουν, στη Λετωνία έκλεισαν λόγω των διώξεων για το ξέπλυμα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πάμε περισσότερο. Φυσικά οι διώξει είναι η λύση. Αν βάλει κανείς στη φυλακή τον υπεύθυνο της KWC ή της Ernst Young όχι ότι έχουν να κάνει κάτι, αλλά άμα τους βάλει κανείς στη φιλική, αν κάνουν κάτι, αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Άμα μπει στη φυλακή ένας δικηγόρος και όχι μόνο ένας τραπεζίτης. Να τους ε, βάλει κανείς στην φυλακή. Αυτό θα ήταν το κατεξοχήν αποτρεπτικό μέσο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγα λεπτά, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Eye δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ο συνεισηγητής μας αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το πάνελ μας. Είναι νομίζω σαφές ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει με το θέμα των χρήσεων θεωρήσεων όπως τις λέμε που είναι το προηγούμενο θέμα αλλά και στο θέμα των ελεύθερων λιμένων. Πρέπει να το δούμε αυτό. Και για μένα είναι σαφές ότι υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα ε, μπορεί να είναι όπως λέει ο κύριος Κάρ ένα ασφαλές μέρος να αποθηκεύσει κανείς ε, τη μαλφή αλλά μπορεί να παραμείνουν εκεί για πάντα, κατά κάποιον τρόπο, και να αλλάζουν οι διοκτήτες χωρίς ε, να υπάρχει επαρκής έλεγχος. Οπότε είναι ένας τρόπος ε, παρανόμου εμπορίου και χρηματικών λόγων. Επίσης, δεν καταλαβαίνουμε τι όφελο ε, έχει αυτό, τι όφελο προσφέρει αυτό το σύστημα για την πραγματική οικονομία. Δεν θεωρώ ότι έχει Οπότε, γνωρίζοντα βεβαίω τα όρια των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Αλλά βεβαίω θα πρέπει η Επιτροπή και εγώ ως εισηγητής να δούμε το ζήτημα. Και πρέπει, όπως είπαν αρκετοί, να είμαστε καλύτεροι όσον αφορά την εποπτεία, την ανείχνευση, αλλά και την, και την δίωξη. και χρειαζόμαστε σαφείς ευρωπαϊκούς κανόνες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας βεβαίως. Είμαστε ειδικά σε μια ένωση όπου υπάρχει ένα άρθρο που λέει ότι πρέπει να υπάρχει ειλικρινή συνεργασία μεταξύ μας για να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα χρήματο κτλ. Ε, εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο λοιπόν. Οπότε το απαιτεί και η συνθήκη πέρα από τις διάφορες οδηγίες ε, περί ξεπλήματος ε, χρήματος. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το πάνελ που μας ε, διαφώτισε σε κάποια ζητήματα και να είστε σίγουροι ότι εμείς θα δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστώ. Γέπε. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώθηκε το πάνελ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις ε, παρεμβάσεις τους ε, και θα ρωτήσω τώρα τους βουλευτές αν έχουν τίποτα στα διάφορα. Όχι, οπότε η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας είναι την 5η 18 Οκτωβρίου στις 2 η ώρα υπό μορφή εργαστηρίου. Σας ευχαριστώ για τη συνεδρίαση.